good afternoon, everybody. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίασή μας. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη εάν δεν έχετε σχόλια. Επόμενο σημείο, έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης 19 και 20 Ιανουαρίου του 2009. Εάν δεν υπάρξουν σχόλια μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης, τα πρακτικά θα θεωρηθούν εγκριθέντα. Στη σημερινή συνεδρίαση θα γίνεται διαδικτυακή μετάδοση, επομένως έχετε την ευκαιρία να αφήσετε το σημάδι σας στην ιονιότητα, για καλό για κακό. Το λέω απλώς για να το γνωρίζετε. Πάμε στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης, προστασία ζωών τη στιγμή της θανάτωσής τους έχουμε τον εισηγητή, τον κύριο Γιάννους Βοησεβόσκη και έχουμε και το θέμα της ανταλλογής απόψεων με εμπειρογνώμονες. Μετά τη συζήτηση τον Ιανουάριο έχουμε προσκαλέσει λοιπόν τέσσερις εμπειρογνώμονες για την ανταλλαγή απόψεων για αυτό το πολύ λεπτό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων και των διαστάσεων της ε, τελετουργικής σφαγής ή της, ε, του σφαγής των ζώων σύμφωνα με ε, τα πρέποντα των θρησκειών. Έχουμε μία ώρα και 40 λεπτά στη διάθεσή μας. Οι εμπειρογνώμονες λοιπόν δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 λεπτά στην παρουσίασή τους και μετά ε, θα ήθελα επίσης και τα μέλη να ζητήσουν το λόγο πριν ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων. Και δεν θα δώσω περισσότερο χρόνο από 10 λεπτά στον καθένα. Στη συνέχεια, ε, οι εμπειρογνώμονες θα επανέλθουν για 3 ή 5 λεπτά για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μελών και ο εισηγητής θα εξάγει τα συμπεράσματα της συζήτησης. Καλωσορίζω θερμά τους εμπειρογνώμονές μας. Τον πρώτο εμπειρογνώμονα, τον κύριο Ζεφ Νόγκα, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίας Ζωικού Κεφαλαίου και Κρέατος. Έχετε το λόγο, έτσι δεν είναι, παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ε, πολύ θερμή πρόσκληση που μου απευθύνετε και θα ήθελα κατά δεύτερο λόγο να σας ε, συστηθώ για άλλη μια φορά. Λέγομαι Ζήιβ Νόγκα, είμαι εκτενίατρος Ισραηλινός με πτυχίο εκτενιατρικής από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και είμαι σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίας Ζωικού Κεφαλαίου και Κρέατος, σύμβουλος κτηνιατρικών θεμάτων. Ως προς την πρόταση κανονισμού για την καλή διαπίωση των ζώων ε, τη στιγμή της φαγής, θα ήθελα να κάνω μια παρουσίαση εστιάζοντας τη θρησκευτική σφαγή και την σήμαση και θα προσεγγίσω ετικετοθεσία, θα προσεγγίσω το θέμα από τρεις σκοπιές, τη σκοπιά της αγοράς, την τεχνική οικονομική σκοπιά, αλλά και τη θρησκευτική σκοπιά. Και ως προς τη θρησκευτική σκοπιά θα παρουσιάσω την προσωπική μου άποψη. Πρώτον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν 29 εκατομμύρια βοηδοί και 72 εκατομμύρια πρόβατα σφαγιάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση κάθε χρόνο. Και το βόλιο και πρόβιο κρέας παράγεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες και κανονισμούς για την καλή διαβίωση, για την δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Όλα τα κρέατα λοιπόν πληρούν τους ίδιους κανόνες και έχουν το, τα ίδια χαρακτηριστικά. Βεβαίως ε, έχουμε θρησκευτικές ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει η βιομηχανία κρέατος να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καταναλωτών. είναι γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σφαγιάζονται ζώα χωρίς αποπληξία. Είναι δύσκολο να ξέρουμε πώς ακριβώς γιατί δεν έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία. Να δούμε το παράδειγμα της Γαλλίας. 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γαλλία ανήκουν στη μουσουλμανική και εβραϊκή κοινότητα. 240.000 τόνοι λοιπόν πρέπει να προχωρήσουν να πάνε στα σφαγεία και τα αντίστοιχα ζώα να σφαγιαστούν χωρίς αποπληξία. Έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ε, βάρος τόνου ε, κουφαριού, το οποίο προκύπτει από ζώα που έχουν σφαγιαστεί χωρίς αποπληξία. Το ίδιο ισχύει και στην ε, σφαγισμό των πουλερικών. Χαρακτηρίζονται λοιπόν όλα αυτά από δύο βασικούς παράγοντες. Το επίπεδο κατανάλωσης είναι γενικότερα υψηλότερο από τον μέσο όρο. Η κατανάλωση εγωπροβάτων στην Γαλλία είναι 8 φορές μεγαλύτερη από, ε, από τον εθνικό μέσο όρο. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, ζήτηση υπάρχει για ορισμένα μέρη των ζώων μόνο. Η η εβραϊκή κοινότητα συνήθως καταναλώνει το εμπρόστατα αρτιμόριο, ενώ η μουσουλμανική κοινότητα καταναλώνει και τα εντόστια και άλλα μέρη του ζώου. Επομένως, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι το εξής. Όλα τα κρέατα που παράγονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωση συμμορφούνται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και έχουν τα ίδια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Το βόλιο και το πρόβιο κρέας το οποίο αποκτάται μέσω της θρησκευτική σφαγής χωρί την τεχνική της αποπληξία, ουσιαστικά είναι ε, μειονότητα στο σύνολο της παραγωγή είναι ένα μικρό κομμάτι και είναι κάτι το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες των θρησκευτικών κοινοτήτων που ενδιαφέρονται για κατανάλωση κρέατος που, ε, ζώων που έχουν σφαγιαστεί χωρίς αποπληξία. Δεύτερο επιχείρημα που θα ήθελα να προβάλλω είναι η μελέτη σκοπιμότητας. Όλες οι, το σχέδιο έκθεσης το ευρωπαϊκό της αντίστοιχης επιτροπής του Κοινοβουλίου βλέπει ότι όλα τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να φέρουν σήμανση. Αυτό λέει το σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη ανάλυση με βάση τις εμπειρίες που έχουμε από το σύστημα σήμανσης στον τομέα του βόηου κρέατος. Αν υποθέσουμε ότι όλα τα προϊόντα θρησκευτική σφαγής θα πρέπει υποχρεωτικώς να φέρουν σήμανση, τότε ο κλάδος θα πρέπει να επιβάλλει σύστημα εχνηλασιμότητας από το σφαγείο μέχρι και τον τελικό καταναλωτή ώστε να αποκτώνται αξιόπιστες πληροφορίες. Το σύστημα λοιπόν της ε, ιχνηλασιμότητας αυτό θα περιλαμβάνει το βόιο, το πρόβιο, ο κρέας αλλά και το κρέας των πουλερικών ζώων που έχουν υποστεί θρησκευτική σφαγή αλλά και των υπολείπων ζώων. Δηλαδή η σήμαση θα είναι ένα ακόμα ε, πληροφοριακό στοιχείο και ίσως αποτελεί και εγγύηση εναντίον της απάτης. Και το σύστημα ποιότητας βασίζεται στην ατομική ταυτοποίηση των ζώων. Αλλά αυτό είναι κάτι που υπάρχει ήδη ως προς τα βοηδή και υπάρχει και στο, ως προς τα ε, εγωπρόβατα. Ωστόσο, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση όλων των προβάτων θα πρέπει να ενοποιηθεί, να παγιωθεί περισσότερο. Έχουμε 96 εκατομμύρια πρόβατα και 30 εκατομμύρια έγες. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα εχνηλασιμότητας ε, πέραν όλων των λάνων να ισχύσει και για τα ε, προϊόντα ε, πρόβιου κρέατος, όπως είναι τα εντόστια για παράδειγμα. Είναι σίγουρα περίπλοκο ένα τέτοιο σύστημα και θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους του κρέατος. Το κόστος της ιχνηλασιμότητας στο βόλιο κρέας αντιστοιχεί σε 330 ε, εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο της ευρωπαϊκής παραγωγής. Και εκτιμάται σε επιπρόσθετη επιβάρυνση 82 εκατομμυρίων ευρώ. Ως προς το πρόβιο κρέας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η επιπρόσθετη επιβάρυνση θα ανέλθει σε 22 εκατομμύρια ευρώ συνολικά 404 εκατομμύρια ευρώ για αυτούς τους τομείς. Βλέπετε λοιπόν ότι η άνοδος του κόστους δεν είναι καθόλου αμεληταία. Εάν ε, λάβει κανείς υπόψη του και το πόσο άκαμπτο, δίσκαμπτο είναι το σύστημα αυτό της χνηλιασιμότητας και σίγουρα θα προκύψουν διάφορες παρενέργειες. Ποιε είναι αυτές. Θα αυξηθεί η τιμή του κρέατος καταρχάς και ειδικότερα τιμή του κρέατος που αγοράζουν οι συγκεκριμένες θρησκευτικέ κοινότητες. Δεύτερον, θα έχουμε παράνομες σφαγές ή ε, σφαγιασμού ζώων εκτός εγκεκριμένων σφαγίων. Ακόμα και στον κλάδο των πουλερικών. Κάτι το οποίο θα υπονομεύσει τη συνολική παραγωγή κρέατος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα έχει και ε, δυσάρεστες συνέπειες και στον οικονομικό τομέα και θα υπονομεύσει κυρίως τις προσπάθειες του νομοθέτη, των παραγωγών, των κρατών, όλων των θεσμικών οργάνων τα οποία μάχονται για να έχουμε ομοιόμορφα νομικά πρότυπα με σεβασμό στην καλή διαβίωση των ζώων, με τήρηση των αρχών δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Το γεγονός παραμένει ότι Μόνο τα ε, κρατικώς επιτηρούμενα σφαγεία είναι σε θέση να εξασφαλίζουν ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Άρα, θα πρέπει αυτό να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Άλλη παρενέργεια ε, θα είναι η αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να επιβάλλει τις ίδιες υποχρεώσεις στις τρίτες χώρες. Νομίζω ότι θα έχουμε μερική αμοιβαιότητα μόνο. Και μόνο τα ε, κρέατα που πολλούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φέρουν σήμανση εάν υιοθετηθεί ε, αυτό το οποίο λέει το σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτι το οποίο θα δώσει μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα στις ε, τρίτες χώρες. Τέλος, ο κλάδος, η βιομηχανία, αυτό το οποίο προτείνει είναι να αφιερώσουμε προσπάθειες στο να εξειδικεύσουμε καλύτερα και να καταρτήσουμε καλύτερα το προσωπικό που εργάζεται, που εργάζεται στα σφαγεία. Και γι' αυτό προτείνουμε αυτή την τροποποίηση στην πρόταση κανονισμού. Η πρόταση ουσιαστικά αγνοεί τις ε, τεχνολογικές προόδους οι οποίες έχουν σημειωθεί. και τις ε, συστάσεις των διαφόρων διεθνών εμπειρογνωμόνων. Καλό θα ήταν να αναθεωρεί τη διάταξη αυτή τρία χρόνια πριν τη λήξη της. Αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη γνώσεων και καλό θα είναι να γίνεται και ενδιάμεση αναθεώρηση. Ένα άλλο συμπέρασμα που θα μπορούσα να εξάγω είναι το εξής. Μία ανάλυση κόστους και ωφέλους δείχνει ότι η σήμανση των προϊόντων ε, σφαγίων χωρίς αποπληξία σύμφωνα με, τις, ε, με τα θρησκευτικά πρότυπα. Είναι κάτι το οποίο αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό προϊόν, αποδυναμώνει την ανταγωνιστικότητά μας και δεν βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων. Η ύπαρξη δηλαδή υποχρεωτική της σήμανσης αυτής. Και θα ήθελα να εκφράσω και την προσωπική μου άποψη. Το, όλο τον προηγούμενο μήνα έχω παρακολουθήσει το θέμα αυτό ε, πολύ προσεκτικά. Έχω συναντηθεί με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της αντίστοιχης Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με εκπροσώπους έχω συναντηθεί επίσης ε, των εβραϊκών και μουσουλμανικών κοινοτήτων αλλά και με διάφορους εμπειρογνώμονες. Ίσως υπάρχει σύγχυση μεταξύ θρησκευτικών αρχών και επιστημονικής γνώσης που προέρχεται από τα διάφορα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα. Το θέμα της καλής διαβίωσης των ζώων τη στιγμή της φαγής είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει ευκρινήσεων. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι μέθοδοι της αποπληξίας που χρησιμοποιούνται. Ο καθένας νομίζω ότι μιλάει από διαφορετική προοπτική. Όσοι στηρίζουν την αποπληξία ε, κατά τη σφαγή προβάλλουν μόνο τα καλά της και τα πλεονεκτήματα και τις μελέτες που μιλούν μόνο για αυτά. Ενώ οι αντίθετοι με την άποψη αυτή εκπροσωπούν μόνο τις δικές τους αρχές, εκφράζουν τις δικές τους αρχές και τονίζουν ότι δεν μπορούν να καταναλώσουν το κρέας με τις ε, μεθόδους, ε, το κρέας που έχει παραχθεί με σφαγή ζώου, με τη μέθοδο της αποπληξίας πριν τη σφαγή. Εγώ προσπάθησα να είμαι αντικειμενικός και να παρουσιάσω ε, την κατάσταση με επιστημονική σοβαρότητα, με βάση την επιστημονική μου την κατάρτιση, αλλά και με βάση την γνώση μου για την εβραϊκή κοινότητα. Κατανοώ πολύ καλά τους φόβους των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη και ε, ξέρετε ότι είναι σημαντικό να τονίσει κανείς ότι οι εβραϊκές κοινότητες έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα και υπάρχουν ακόμα στην Ευρώπη ακριβώς διότι έχουν σεβαστεί τις ε, αρχές ε, της βίβλου τους χωρίς να παρεκκλίνουν από τις αρχές τους κατά την ε, πάροδο των αιώνων. Και Εάν αλλάξει έστω και ένας κανόνας σε αυτό το στάδιο, αυτό το ε, αντιμετωπίζουν οι κοινότητες οι εβραϊκές ως απειλή στο συνολικό τρόπο ζωής τους. Θεωρούν ότι αυτό είναι πραγματική απειλή στη θρησκεία τους. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό και με βάση τις αρχές της επιστήμης αλλά και με βάση τις αρχές της συνείδησής σας. Ευχαριστώ. Ναι, θα το εξετάσουμε και κατά συνείδηση και λαμβάνοντας υπόψη μας ε, την ε, επιστήμη. Ε, ο επόμενος ομιλητής είναι ο ε, Ραβίνος και εκτινίατρος. Ε, σας παρακαλώ ε, να προσπαθήσετε να παραμείνετε εντός των χρονικών ορίων. Εκτός μικροφώνου ο ομιλητής. Je sais pas, il marche. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Είμαι ο Ραβίνος Φίζο. Ε, και είμαι επίσης και εκτίνοτρόφος, ε, κάτι το οποίο εξηγεί κάπως ε, την παρουσία μου εδώ. Θα ήθελα να πω και μερικά πράγματα στα αγγλικά, να σας πω ποια είναι και η εβραϊκή θέση. Ο σφαγιασμός δεν μπορεί να είναι... Ε, κάτι το ανθρώπινο ε, υπό καμία, σε καμία περίπτωση, αλλά μπορεί να γίνει με όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινο τρόπο. Αυτή είναι η θέση ε, η εβραϊκή. Γνωρίζουμε ότι τώρα η βίβλος ε, μας ε, ζητά να μην κάνουμε τα ζώα να υποφέρουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες, ε, ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο και γι' αυτό προσπαθήσω να τον σεβαστώ. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί κανόνες που επιτρέπουν την ευημερία των ζώων και αυτός που σφαγιάζει το ζώο έχει πολύ μεγάλη ευθύνη όσον αφορά τον περιορισμό του πόνου του ζώου. Να σκεφτούμε τώρα μερικά ζητήματα νομικά. Καταρχάς, ε, η αναισθησία είναι κάτι το πάρα πολύ ε, σημαντικό. Αν δεν το λαμβάνουμε υπόψη, ερχόμαστε σε αντίθεση με απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι η τελετουργική σφαγή είναι ένα σημαντικό ε, είναι μια σημαντική πτυχή που δίνει τη δυνατότητα της ασκήση της ελευθερίας ε, ε, των θρησκειών με το με, του άρθρου 9 των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρόκειται λοιπόν για ένα τυπικό, ένα τελετουργικό, στο οποίο είμαστε πάρα πολύ αφοσιωμένοι και μάλιστα και το βελγικό κράτος, δεν θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες, έχει σχετική απόφαση όσον αφορά την κυρία Γιώ Μαρή ε, είχε αποστείλει μία επιστολή προς τον πρόεδρο Μπαρόσο και είχε πει ότι αυτές οι θεμελιώδεις ελευθερίες είναι μία, ένα κεκτημένο των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως όπως αναφέρει άλλωστε και η συνθήκη της Λισαβόνας. Τα πράγματα λοιπόν είναι τελείως σαφή. Τώρα να δούμε τι ακριβώς σημαίνει το τυπικό, ο σφαγιασμός, ο τελετουργικός σφαγιασμός. Πρέπει να είναι υγιές το ζώο και να μην υπάρχουν ε, πληγές. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς δεν θέλουμε ε, την ε, αναισθησία προηγουμένως. Γιατί ακριβώς, θα γίνω λίγο τεχνικός γιατί είναι σημαντικό για τη συζήτηση, πρέπει να κόψουν βέβαια την καροτίδα και διάφορα μέρη του ζώου δεν, ε, δεν όμως δεν πλήττονται τα πολύ κέρια όργανα όμως του ζώου, ε, δηλαδή αυτός που σφαγιάζει έχει μία πάρα πολύ καλή εκπαίδευση γιατί ε, γιατί ακριβώς ε, πρέπει όσο το δυνατόν ε, πιο καλά να λάβει υπόψη του τον περιορισμό του πόνου του ζώου. Υπάρχουν και σχετικές επιστημονικές μελέτες, υπάρχουν και αποτυχίες της αναισθησίας σε 6,5% των περιπτώσεων, επομένως τα αριθμητικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Πρόκειται για κάτι το οποίο αναφέρει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, για το οποίο θα επανέλθω αργότερα. Όταν μιλάμε τώρα για κοπή τη καροτίδα, ε, μειώνεται πάρα πολύ η πίεση ε, του αίματο του ζώου, ε, υπάρχει ισχυμία των νευρικών κυτάρων, δεν τροφοδοτούνται, δεν τροφοδοτούνται πια για, 5 έως, για 0 έως 5 δευτερόλεπτα. Πέφτει πάρα πολύ η πίεση στις αρτηρίες. Όσον αφορά την αρτηρία όμως η οποία ε, βρίσκεται στη σπονδυλική στήλη και η οποία δεν κόβεται. Αυτή η τροφοδοσία γίνεται σε πολύ, είναι, είναι πλέον πολύ μικρή, αυτή στιγμή ε, κόβεται και επομένως ε, η μείωση της πίεσης σε αυτή την αρτηρία είναι αρκετά σημαντική. Τώρα, το εγκεφαλογράφημα, το πόσο δηλαδή λειτουργεί ο εγκέφαλος και αυτό δείχνει πόσο έχει ε, συνέστηση το ζώο. είναι ο λιγότερο κακός ε, τρόπος τέλος πάντων για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο υποφέρει το ζώο και κατά πόσο έχει συνείδηση του τι συμβαίνει. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω εξέταση. Τώρα όσον αφορά την έκθεση για τα ε, εγκεφαλογραφήματα ε, γνωρίζετε και τους σχετικούς πίνακες, τους έχετε στη διάθεσή σας, μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι ότι το ίμιση της τροφοδοσίας του εγκεφάλου με, ε, με μηνύματα ε, επιτυγχάνεται πιο ε, καλά με το τυπικό τελετουργικό. Αυτό αποδεικνύεται. Αυτό που δημιουργεί προβλήματα και αυτό Αφορά βέβαια κάποιες περιπτώσεις, ε, σε μερικές τέλο πάντων περιπτώσεις συγκεκριμένων ζώων. Ε, ένα ζώο μπορεί να χρειαστεί 60 με 80 δευτερόλεπτα για να χάσει την, ε, τις αισθήσει του. Αλλά αυτό είναι μια πάρα πολύ εξαιρετική περίπτωση. Όσον αφορά τώρα τα επιστημονικά στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες οι οποίες ε, ουσιαστικά οδηγούν ε, σε ισοδυναμία του τελετουργικού σφαγιασμού σε σχέση με τις άλλες μεθόδους ε, σφαγιασμού κατόπιν αναισθησίας, αποπληξίας κλπ. Δεν θα μιλήσω τώρα για το γεγονός ότι όταν κόβεται ο λαιμό των ζώων δεν έχουν συνέστηση τα ζώα. Είναι τόσο ελάχιστο το χρονικό διάστημα που δεν έχουν αίσθηση. Και μάλιστα αναφέρεται ότι είναι και μία τελείως ανώδυνη μέθοδος σφαγιασμού των ζώων. Αυτό αναφέρεται από σημαντικούς καθηγητές και εμπειρογνώμονες. Δεν πρέπει να γύρει πλάστιγκα προς τη μία ή την άλλη ε, μεριά. Ο κτηνίατρος ε, ε, Μπενιντζέρ, καθηγητής κτηνιατρικής στο Παρίσι, ανέφερε ότι παλαιότερα βέβαια όσον αφορά το τελετουργικό σφαγιασμό έλεγε ότι το γεγονός ότι αυτό αποτελεί σκληρό τρόπο σφαγιασμού δεν αποδεικνύεται επιστημονικός. Και άλλες τέτοιες μαρτυρίες υπάρχουν ότι όταν υπάρχει αναισθησία προηγουμένως, ε, η σημασία για την ευημερία των ζώων δεν αποδεικνύεται. Ειδικότερα αν λάβουμε υπόψη ε, το πόσο σημαντικό, πόσο σημαντικός είναι ο πόνος ε, που νιώθουν τα ζώα στα προηγούμενα στάδια του σφαγιασμού όταν υπάρχει αναισθησία για παράδειγμα. Γι' αυτό θα θέσουμε το θέμα που μας δημιουργεί μας πρόβλημα. Καταρχάς, το θέμα ε, ε, των παρεκκλήσεων. Ε, για παράδειγμα, η οδηγία σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησία, αλλά, όλες, ε, αλλά πάντοτε μπορεί να υπάρχει μία εξαίρεση. Όλα τα κράτη-μέλη δηλαδή μπορούν να αποφασίσουν ε, να ε, δώσουν εξαιρέσεις. Είναι μια πρακτική που ήδη υπάρχει και μάλιστα ε, μιλάω κυρίως για χώρες ε, στις οποίες ε, υπάρχουν πολιτικές πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για το σφαγιασμό του ζώου όταν είναι όρθιο. Αυτό ε, απαγορεύεται. Και βασιζόμαστε σε μια έκθεση της ΕΦΣΑ μάλιστα που συγκρίνει αυτό το σφαγιασμό όταν το ζώο είναι όρθιο στο ε, κουτί περιορισμού, στο κυβότιο περιορισμού του ζώου πριν από το θάνατό του και θεωρεί ότι είναι παροχημένο, ότι δεν χρησιμοποιείται όχι, πλέον γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και προτιμούμε το σφαγιασμό του ζώου ε, χωρίς να είναι όρθιο. Και δεν ε, εννοούμε βέβαια ότι δεν είμαστε υπέρ της ευημερίας των ζώων. Ε, ε, δεν, διαφωνούμε με την ευθύνη όσων σφαγιάζουν τα ζώα των υπευθύνων σφαγής και βέβαια Σύμφωνα με τον κύριο Εντσέρ, ε, εμπειρογνώμονα της ε, ΕΕΦΣΑ, δεν ε, υπάρχει κανένας, κανένα επιπλέον όφελος όταν το ζώο σφαγιάζεται όρθιο. Τώρα, όσον αφορά την ετικετοθεσία, κάτι το οποίο πραγματικά θα δημιουργούσε πρόβλημα στους, στην εβραϊκή και μουσουλμανική κοινότητα, γιατί θα έθετε να αμφιβόλω όλο το σύστημα παραγωγής. Ο κύριος Μπαρνιέ είχε ήδη ε, εκφράσει την άποψή του ως προς αυτό. Εμείς, ε, εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα αυτό, γιατί οι πληθυσμοί η εβραϊκή και η μουσουλμανική της Ευρώπης, ναι βεβαίως θέλουν να συμμετάσχουν ε, σε αυτήν την ευρωπαϊκή οικονόμηση, αλλά δεν πρέπει να είναι και ένα ιδιωτικό θέμα στο οποίο οι Εβραίοι και οι μουσουλμάνοι δεν θα μπορούν να ζουν, γιατί δεν θα μπορούν να ασκούν τις βασικές τους ελευθερίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο γιατρός Αρκάντα Άπη, ημάμ της Λίον, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου άποψη για τα θέματα αυτά, αλλά και την άποψη του ε, Προέδρου του Γαλλικού Μουσουλμανικού Συμβουλίου και του θεσμικού ε, οργάνου εκπροσώπησης μουσουλμανικής κοινότητας στις κάτω χώρες. Θα ήθελα καταρχάς να σας εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες για την ακρόαση που μας έχετε επιφυλάξει στο πλαίσιο της, ε, των εργασιών σας για το θέμα αυτό το πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Θέλω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας τις ανησυχίες μας. Δεν ε, ξεκινήσατε χθες να δουλεύετε για αυτό το θέμα, όμως ε, δεν έχετε ε, λάβει υπόψη σας, δεν έχετε ζητήσει τη συμμετοχή των θρησκευτικών κοινοτήτων. Ίσως θεωρήσατε ότι θα παραμείνει το status quo έτσι όπως έχει ως προς την θρησκευτική σφαγή. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Το άρθρο 4 του σχεδίου κανονισμού θα αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση, το καθεστώς που ισχύει αυτή τη στιγμή για την θρησκευτική σφαγή, αλλά θα πλήξει και άλλες αρχές οι οποίες θυσιάζονται στο, στο βωμό της ε, έλλειψης ανεξιθρησκείας θα έλεγα και στα 10 λεπτά που μας δίνετε κύριε Πρόεδρε θα προσπαθήσω να διευκρινίσω και να επισημάνω τα πιο σημαντικά για μας ζητήματα. Η μουσουλμανική θρησκευτική σφαγή είναι μία βασική αρχή για μας διότι βασίζεται η αρχή αυτή στην έννοια του νομίμου και του παρανόμου σύμφωνα με τις ε, μουσουλμανικές επιταγές. Μιλώ για την αρχή της ε, προφύλαξης και αναφέρομαι πάντοτε στο άρθρο 4. Και ε, μια άλλη αρχή η οποία έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική και είναι η αρχή της επικουρικότητας. Θέλω λοιπόν να επικαλεστώ την αρχή της ε, προφύλαξης και την αρχή της επικουρικότητας για να υπερασπιστώ τα επιχειρήματά μας. Υποτίθεται ότι θέλουμε να βοηθήσουμε στην καλή διαβίωση των ζώων. Όμως ε, για να το κάνουμε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ουσιαστικά ισλαμοφοβική και πάρα πολύ δογματική. Η θρησκευτική σφαγή προστατεύεται ε, από διάφορα κείμενα, από κείμενα που έχουν να κάνουν όπως είναι ας πούμε οι συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τους Υπουργούς της 17 ε, Ιανουαρίου του 2001, ε, από κείμενα όπως η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και άλλα νομοθετήματα, πληθώρα νομοθετημάτων απαλλάσσουν ε, την θρησκευτική σφαγή. Η μοναδική παρέκκληση είναι η παρέκκληση που δίδεται στην θρησκευτική σφαγή. Και δίδεται αυτή η παρέκκληση ακριβώς εξ ονόματος των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο έχουμε εγγράψει στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μιλώ βεβαίως για το δικαίωμα ε, της, ε, του ελευθερώ ασκήν μια θρησκεία και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την αρχή της προφύλαξης την οποία ανέφερα και στην αρχή. Ε, λέει λοιπόν η μουσουλμανική θρησκεία ότι είναι σαφώς καθορισμένα τα πεδία του νομίμου και του παρανόμου. Υπάρχουν όμως κάποιες καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να απομονωθούν γιατί μπορεί να μετακυλήσουν στο μέλλον προς την άλλη κατεύθυνση. Και εδώ είναι που εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης. Βεβαίως το Ισλάμ απαγορεύει την, ε, τον βασανισμό των ζώων ή την ε, χρήση, χρησιμοποίηση των ζώων για λόγους ψυχαγωγίας, όπως είναι η ταυρομαχίας για παράδειγμα. Οποιοδήποτε θύραμα ε, έχει βληθεί με βλήμα δεν μπορεί να καταναλωθεί, διότι υπάρχει αμφιβολία για το πώς πέθανε το ζώο αυτό. Ε, πέθανε επειδή δέχτηκε το βλήμα ή πέθανε επειδή πυροβολήθηκε από τον κυνηγό και κατέληξε σε ένα ριάκι σε μια λίμνη και τελικά πνιγήκε. Βλέπετε ότι ο Ισλάμ προβλέπει όλες αυτές τις αρχές και γι' αυτό είμαστε κατά της ε, αποπληξίας εκ των υστέρων μετά τη σφαγή αλλά και της ε, και όλων αυτών των ε, πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και η OIE το μόνο που λένε είναι ότι δεν υπάρχει ε, αξιόπιστη μέθοδος αντιστρέψιμης παποπληξίας η οποία να εγγυάται 100% την ε, εκ την αναβίωση αν θέλετε του ζώου. έχουν υιοθετηθεί διάφορα ψηφίσματα σε παγκόσμιο επίπεδο για την, για την καλή διαβίωση των ζώων. Πιο συγκεκριμένα υιοθετήθηκαν αυτά στις 20 και 22 Οκτωβρίου στην διάσκεψη του Καΐρου στην, Αίγυπτο και δεν θα πρέπει να τα λησμονούμε διότι ο ΑΗ θεωρεί ότι με δημοκρατικό και διαφανή τρόπο θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι αρχές οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται στην δεοντολογία, την ηθική αλλά και στις επιστημονικές γνώσεις λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, περιφερειακά, πολιτισμικά, ε, πολιτιστικά, ε, θρησκευτικά ε, θέματα, πτυχές και διαστάσεις δηλαδή το άρθρο 4 έτσι όπως έχει συνταχθεί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά προσβάλλει ε, την ε, αρχή της ανεξιθρησκείας. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν αυτή την προστασία με αποτελεσματικό τρόπο, διότι η θρησκευτική ελευθερία είναι θεμελιώδης ελευθερία. η διατήρηση της θρησκευτική σφαγής είναι κάτι το πολύ ε, σημαντικό. Δηλαδή η απουσία εκ των προτέρων αποπληξίας. μπορούμε να εκχωρήσουμε την, ε, ε, το, τη δυνατότητα αυτή στις τοπικές αρχές να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της επικορικότητας. Δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι, πού θα πρέπει να απευθυνθούν για να διεκδικήσουν αυτή τη θρησκευτική τους ελευθερία. Εάν ε, όλα τα κράτη-μέλη αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να εφαρμόσουν την παρέκκληση που έχει δοθεί, να επιτρέπεται δηλαδή η θρησκευτική σφαγή, δηλαδή να μην γίνεται αποπληξία πριν τη σφαγή. Πού θα αποτανθούν, σε ποιον θα στραφούν όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτες. υποτίθεται ότι ε, εκπροσωπείτε αυτούς που σας έχουν εκλέξει. Ε, σας καλώ να συμβουλευτείτε τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε πάρα πολλές γραπτές ερωτήσεις. Έχουμε γραπτή ερώτηση από τον βουλευτή Μουσκαρντίνη στις 20 Ιανουαρίου του 2009 και περιμένω την απάντηση. Είναι πολύ λυπηρό να διαπιστώνει κανείς ότι ακόμα και στους κόλπους του Κοινοβουλίου υπάρχει αυτή η αιμονή ε, να χαρακτηρίζεται η θρησκευτική σφαγή ως μια πράξη βάρβαρη και χαρακτηρίζεται με απαράδεκτους επιθετικούς προοριζορισμούς θα έλεγα. Άλλες ερωτήσεις άλλων βουλευτών ουσιαστικά αποτελούν ε, κερδοσκοπική προσέγγιση των ε, στατιστικών στοιχείων και αριθμητικών στοιχείων. Ζητούμε λοιπόν τροποποίηση του άρθρου 4. Δεν θα επανέλθω σε όλα αυτά τα οποία είπαν πολύ σωστά ο κύριος Νόγκα και ο κύριος Φιζόν. Ε, θα έλεγα όμως ότι η υποχρέωση σήμασης είναι μια ιδέα που φαίνεται καλή, αλλά ουσιαστικά είναι λάθος, είναι εσφαλμένη. Μια, ένα τέτοιο σύστημα σήμασης είναι, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα αρκετά περίπλοκο. Καταρχάς, κρέας που προέρχεται από ζώο που δεν έχει υποστεί αποπληξία δεν έχει διαφορετικά οργανοληπτικά ή διατροφικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά από το άλλο. Ο έλεγχος της σήμασης είναι αδύνατος. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική δοκιμασία, ένα τεστ που να επιβεβαιώνει ότι αυτός που φέρει σήμανση ε, έχει εκπληρώσει τον κανόνα που προβλέπεται. Τρίτον, δεν γίνεται να εφαρμοστούν οι ίδιες οι ίδιοι κανόνες στις τρίτες χώρες. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εθνοτική σήμανση η οποία θα στιγματίσει τις κοινότητες την εβραϊκή και τη μουσουλμανική είναι μια σήμανση εθνοτικού χαρακτήρα και θα ε, βλάψει την αγορά και αντιβαίνει στις ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπερασματικά κυρίες και κύριοι, ελπίζω ότι έχω συμβάλει στον προβληματισμό σας, στην, ε, ε, στην επεξεργασία αυτών των θεμάτων και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε περισσότερες ερωτήσεις. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Δόκτωρ Μισελ Κοράτ από την Eurogroup. Είσαστε και εσείς κτηνίατρος και εμπειρογνώμων στη σφαγή. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συστηθώ σύντομα. Όπως είπατε είμαι μεγάλος κτηνίατρος και εργάζομαι για την Eurogroup εδώ και ένα χρόνο. Πριν από αυτό όμως, 9 χρόνια πέρασα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως επίσημος κτηνίατρος, εργαζόμενος ε, σε σφαγεία στην αρχή της παρέμβασής μου. Θα ήθελα να πω σαφώς ότι ως ε, οργάνωση προστασίας των ζώων δεν είμαστε κατά των, της θρησκευτική σφαγής, είμαστε κατά της ε, σφαγής ε, χωρίς ε, προηγούμενη αναισθητοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. κάποια νούμερα έδωσε ο, ο Νούγια, αλλά είναι ένα θέμα που ξεπερνάει το, το θρησκευτικό τομέα. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο τα τελευταία στοιχεία της κυβέρνησης λέγανε ότι το 2005 το 92% των ε, προβάτων ε, σκοτώθηκαν χωρίς ε, προηγούμενη αναισθητοποίηση. 92% η θρησκευτική κοινότητα είναι πολύ μικρότερη από αυτά. Αν πάρουμε τα γαλλικά στοιχεία, τα αντίστοιχα νούμερα είναι το 40% των αγελάδων, 25% των μοσχαριών και περίπου το 55% των προβάτων που στη Γαλλία σκοτώνονται διαμορφώνονται χωρίς ε, προηγούμενη αναισθητοποίηση. 8% όμως ε, είναι ο μουσουλμανικός και εβραϊκός ε, πληθυσμός. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη διαφορά στα νούμερα. Να αναφέρω ποια είναι η κατάσταση του θέματος αυτού της θρησκευτικής φαγής σε όλο τον κόσμο, διότι νομίζω ότι θα μάθουμε πολλά από αυτό. ακούσαμε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τους συναδέλφους. Ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, στην Ευρώπη Έχουμε κάποιες ε, χώρες όπου απαγορεύεται ε, η ε, σφαγή χωρίς προηγούμενη αριστοποίηση, Νορβηγία, Σουηδία και Ελβετία ε, αναισθητοποίηση όμως αμέσως μετά την, το κόψιμο της ε, ε, σε, περίπτωση που έχει σκοτωθεί ε, ζώο χωρίς ε, αναισθητοποίηση. Ε, αυτό ε, επιτρέπεται σε χώρες, στη, Αυστρία, την Εστονία και την Σλοβακία. Ας μην ξεχνάμε ότι η Φιλανδία και η Δανία έχουν περιορισμένα μέτρα τέτοιου τύπου. Στη Γερμανία έχουμε μια ενδιαφέρουσα κατάσταση, περιορίζεται η σφαγή των ζώων ε, σε, ε, σε πελάτες ε, της θρησκείας αυτής. Επιλέγονται λοιπόν πριν τη σφαγή τα ζώα ανάλογα με τους αναμενόμενους πελάτες. Στον υπόλοιπο κόσμο ε, έχουμε πολύ σημαντικές χώρες που επιτρέπουν την ανιστοποίηση μετά το κόψιμο της ε, καροτίδας σε περίπτωση που δεν έχει ανιστοποιηθεί το ζώο πριν από αυτό. Έχουμε την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Νότια Αφρική. Μεγάλες χώρες ε, λοιπόν έχουν εισάγει το μέτρο αυτό της εκ των υστέρων Κάποιες από τις χώρες αυτές εφαρμόζουν το μέτρο αυτό εδώ και δεκαετίες. Πιο πολύ όμως εκπλήσει το γεγονό ότι κάποιε άλλες χώρες επιτρέπουν τη θρησκευτική σφαγή και αναισθητοποίηση ταυτόχρονα, διότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η θρησκευτική σφαγή δεν ε, σημαίνει ε, σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση. Ε, στην Ναμίμπια, την Συρία, την Ουγκάντα, την Κένια και άλλες χώρες ε, τα ζώνες αισθητοποιούνται πριν την σφαγή τύπου χαλάλ. Σε χώρες όπως ε, η Μαλαισία εισάγονται κρέατα από την Αυστραλία και ε, απέτηση στην Αυστραλία είναι εκ των πριτέρων ε, ε, αναισθητοποίηση και επίσης έχουμε την Γιορδανία όπου έχουμε τεχνικές προηγούμενης αναισθητοποίησης λόγω των προσπαθειών της πριγκίπισσας της χώρας. Έχουμε όμως και τη μη, μη, τις μεθόδους αναισθητοποίησης με μη διατριτική ράβδο. Ε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ε, Ευρώπη έχουμε κάποιες ε, μεθόδους εκ των υστέρων αναισθητοποίησης. Κάποια σφαγεία στην Αγγλία, σφαγεία που σφάζουν κρέατα κόσερ, Έχουμε εκ των υστέρων αναισθητοποίηση που αναφέρεται ρητά στην Υπουργική Έκθεση. Επίσης κάποιες κοινότητες εφαρμόζουν την εκ των υστέρων αναισθητοποίηση ε, και στην Ευρώπη σε πάρα πολλά σφαγεία πουλερικών χρησιμοποιείται η ηλεκτρική αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή. Ας ε, μιλήσουμε τώρα για το γιατί σφάζονται τα ζώα χωρίς αναισθητοποίηση. Ε, αυτό συμβαίνει για θρησκευτικούς λόγους και θα επανέλθω στο θέμα αυτό που εξήγησαν οι συνάδελφοι. Θέλουν τα ζώα να είναι ζωντανά και με ε, στηριακή αντίληψη κατά τη στιγμή της ε, σφαγής. Ε, υπάρχει όμως και εμπορικός λόγος. Γιατί θέλει η ε, βιομηχανία κρέατος να σφάζει χωρίς ανιστοποίηση επειδή είναι πιο, πιο γρήγορο, πιο φτηνό, ε, ένα πρόσωπο λιγότερο στην αλυσίδα παραγωγής και μπορεί και δύο ή τρεις ε, εργαζόμενους λιγότερο και ο δόκτωρ που μίλησε πριν το ανέφερε αυτό. Εάν δεν ανιστοποιηθεί το ζώο, τότε... Ολόκληρο το ζώο θεωρείται ότι έχει σφαγεί με θρησκευτικό τρόπο. Ε, πρόκειται για σημαντική αγορά αυτή που ε, απευθύνεται σε ε, μουσουλμάνους. Η βιομηχανία κρέατος λοιπόν έχει οικονομικά κίνητρα να σκοτώνει χωρίς προηγούμενη ανιστοποίηση. Άλλος λόγος είναι ότι έτσι έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν σε διάφορες αγορές. Τα ζώα που έχουν σφαγεί χωρίς αναισθητοποίηση μπορούν να εξαχθούν ε, σε πολλές αγορές. Επίσης υπάρχουν πολιτικοί λόγοι. Στο παρελθόν υπήρχε σαφής πίεση στους πολιτικούς να μην παρεμβαίνουν σε θρησκευτικά ζητήματα. Οι πολιτικοί συχνά φοβούνται τις ε, ε, Αντιδράσει των ε, θρησκευτικών ε, αρχών και επίσης ε, πίεση ασκεί και η βιομηχανία κρέατος, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Είναι πολύ σημαντικό το λόμπι της βιομηχανία κρέατος. Σας παρουσίασα τα γεγονότα. Υπάρχει λοιπόν λύση στο πρόβλημά μας. Όλοι εδώ πέρα έχουμε κάτι κοινό. Θέλουμε να προωθήσουμε την προστασία των ζώων. Υπάρχει λοιπόν λύση. Άκουσα δύο συναδέλφους που είπαν ότι δεν ε, είναι αποδεκτή η αναισθητοποίηση μετά ε, το κόψιμο της καροτίδας. Ε. Για διάφορους λόγους. Λένε ότι δεν είναι χρήσιμο, δεν έχει νόημα. Είναι δυνατό να γίνει αυτό, όμως η αναισθητοποίηση εκ των υστέρων έχει διάφορα πλεονεκτήματα. Αυτό σημαίνει ότι το ζώο αναισθητοποιείται αμέσως μετά την, το κόψιμο της καροτίδας. Στην ε, Αυστραλία αυτό γίνεται αμέσως κατά τη σφαγή, ε, ενώ στην Νότια Αφρική έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των θρησκευτικών ε, αρχών και θα μας απαντήσουν σε αυτό, αλλά το ζώο φτάνει ζωντανό, υγιές και με διακή αντίληψη κατά την αφέβαση, κατά το κόψιμο της καροτίδας. το ζώο θα αφαιμαχθεί τελείως. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι τα ζώα που αναισθητοποιούνται δεν χάνουν λιγότερο αίμα από αυτά που δεν έχουν αναισθητοποιηθεί. Η αφέμαξη λοιπόν θα είναι ε, εξίσου πλήρης και στις δύο περιπτώσεις. Είναι μέθοδος που σέβεται την προστασία του ζώου δεν ε, ε, πονάει επιπλέον το ζώο διότι ε, ήδη έχει χάσει την ευαισθησία του. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν μπορούμε να αναισθητοποιήσουμε το ζώο με τον τρόπο αυτό. Για σας δεν αλλάζει τίποτα, διότι έχει ήδη αναισθητοποιηθεί το ζώο. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. τώρα ας μιλήσουμε για τους εμπορικούς ε, παράγοντες. τι αλλάζει εδώ. για τα βοηδή. ο χρόνος αφέμαξης είναι αρκετά λεπτά για τα βόηδη. Εάν χρησιμοποιεί κανείς ανεστοποίηση εκ των, εκ των υστέρων, ε, μπορεί να μειωθεί ο χρόνος σε 30 δευτερόλεπτα. Για εμπορικούς λόγους λοιπόν ε, θα εξοικονομηθεί πολύ χρόνος. Ε, ε, έτσι λοιπόν πρόκειται για εξοικονόμηση χρήματος. Για τα πρόβατα δεν αλλάζει τίποτα για λόγους ε, υγείας και ασφάλειας είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνο ε, στα σφαγεία να ε, ανεστοποιούνται τα ζώα διότι δεν κλωτσάνε, δεν, κινού, δεν, δεν κουνιούνται κλπ. Από ε, Γάλλους φορείς εκμετάλλευσης λοιπόν μας λένε ότι είναι δύσκολο για αυτούς να παρακολουθούν ένα ζώο για 2, 3, 4 λεπτά να κινείται μέχρι να κινητοποιηθεί τελείως. Λοιπόν, οι, οι θρησκευτικέ αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης, ε, εμείς ε, που είμαστε οργάνωση προστασίας ε, των ζώων, μπορούμε να δεχτούμε τη λύση αυτή και δεν είναι καλή λύση, είναι απλά καλύτερη λύση από την προηγούμενη, διότι μειώνει τον χρόνο ευαισθησίας του ζώου. Έλαβα email από τον Δόκτωρα ε, και μου απάντησε ότι ε, η εκ των υστέρων ανιστοποίηση μειώνει το χρόνο ευαισθησίας ε, του ζώου. Το ζώο δηλαδή δεν έχει χάσει τελείως αισθηριακή αντίληψη και ευαισθησία, αλλά ο χρόνος ε, πόνου μειώνεται. Και τέλος, γιατί η πολιτική θα είναι ικανοποιημένη με μια τέτοια λύση, διότι μια και καλή θα μπορέσουμε να σταματήσουμε να μιλάμε για θέματα ε, θρησκευτική φαγής. Εάν μπορέσουμε να συμβαστούμε ε, με τη λύση της ε, εκ των υστέρων ανιστοποίησης αμέσως μετά το κόψιμο της καροτίδας ε, θα είναι ε, ικανοποιητική λύση για όλους. Δεν λέω ότι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι αλλά πιστεύω ότι όλοι θα μπορέσουμε να θεωρήσουν αποδεκτό τον τρόπο αυτόν. έχω και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε νομίζω όμως ότι πρέπει να περάσουμε στη συζήτηση. το μόνο που θα πω ακόμα είναι ότι έχουμε μία πιθανή λύση. Ε, άλλες μεγάλες χώρες, η Αυστραλία, η Νότια Αφρική, η Αυστρία στην Ευρώπη ήδη έχουν επιλέξει ε, την μέθοδο αυτή. Σας παρακαλώ μην χάσετε την ευκαιρία αυτή να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο Ζώσεφ Τόλ μόλι ήρθε, καλώ ήρθε. Ε, Πολλοί από εσά θα τον ξέρετε, ήταν ε, πρώην πρόεδρο ε, τη Επιτροπή Γεωργία. Έχω εδώ ένα κατάλογο των ομιλητών. Προτού να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να πω σαφώ ότι εδώ σήμερα δεν συζητάμε τη θρησκευτική σφαγή και τις ηθικές ε, ούτε προσπαθούμε να επιβάλλουμε τους κανόνες μας και τους νόμους μας σε εσά. Γνωρίζουμε όμω ότι υπάρχει ένα θέμα προστασία των ζώων, ευζοία των και σε περίπτωση που εκτρέφονται ζώα και σφάζονται, εμείς ε, οι άνθρωποι επιλέγουμε πώς σφάζονται τα ζώα αυτά. Πρόκειται λοιπόν για μια πραγματική συζήτηση για να δούμε ε, αν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε. Πολλοί από εμά πιστεύουμε ότι υπάρχει πόνος χωρίς αναισθητοποίηση του ζώου, τελεπορείται το ζώο. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε ε, μια μερική αναισθητοποίηση εκ των προτέρων πριν τη σφαγή ή αμέσως μετά την σφαγή ε, Περί αυτού πρόκειται η συζήτηση σήμερα. Δεν, ε, θέλω όμως να τονίσω ότι δεν καταδικάζουμε καμία θρησκεία, δεν είναι αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που με ξέρουν, ξέρουν πόσο ε, ισχυρέ είναι οι θέσει μου για το θέμα αυτό, για το θέμα της προστασίας των ζώων. Δεν έχει λοιπόν να κάνει με καμία θρησκεία το θέμα, έχει να κάνει με το πώ φάζουμε τα ζώα μας ε, στην Ευρώπη. Κύριε Βόιτσεχόφσκι, θέλετε να ε, παρέμβετε, άλλωστε εκπονείτε την έκθεση αυτή για την Επιτροπή Γεωργίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Όταν αποφάσισα να βοηθήσω στη σύνταξη αυτής της έκθεσης, ήξερα ότι το κείμενο δεν θα ήταν καθόλου εύκολο. Τα ζητήματα είναι πολύ λεπτά, πολύ ακαθόδη. Είναι ένα εξαιρετικό δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Και αυτό που θα ήθελα να πω καταρχάς είναι το εξής. Όταν ε, συνέταξα το σχέδιο έκθεσης, ε, προσπάθησα να προσεγγίσω το ζήτημα που, πάνω στο οποίο θέλουμε να νομοθετήσουμε, ε, σεβόμενος αμφότερες θρησκευτικέ κοινότητες θρησκευτικέ κοινότητε, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα και οι οποίες εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Ενδιαφέρονται ιδιαίτερω για το θέμα αυτό και λογικό. Θέλω λοιπόν να πω εξ αρχή το εξή: Ούτε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε το σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, δεν έχουν σκοπό να περιορίσουν ε, τα θρησκευτικά δικαιώματα. Άλλωστε η θρησκευτική σφαγή θα είναι παρούσα στην πολωνική νομοθεσία και θα συνεχίζει να είναι δυνατή. Δεν συζητούμε δηλαδή το κατά πόσο θα παγορεύσουμε ή θα επιτρέψουμε τη θρησκευτική σφαγή. Ε, προσπαθούμε να προβάλλουμε μία πρόταση συμβιβασμού, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κοινότητες, πάρα πολλοί κύκλοι ανθρώπων, πάρα πολλές ομάδες που θέλουν να εφαρμοστεί μια τέτοιου είδους απαγόρευση. Δεν είναι σωστό λοιπόν να μιλούμε για, ανεξιθρησκεία, για έλλειψη ανεξιθρησκείας και για διακρίσεις εις βάρος τεινός. Ουσιαστικά ε, πολύ συχνά γίνεται λόγος για ε, τρόπο φαγής ο οποίος προκαλεί περισσότερη οδύνη στα ζώα από ότι κάποιος άλλος τρόπος σφαγής. Εξού και προέκυψε η πρόταση περιορισμού των μεθόδων, περιορισμού δηλαδή της θρησκευτικής φαγής ή έστω και απαγόρευσης αυτής. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός μας. Δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε την θρησκευτική σφαγή και θέλω αυτό να το καταστήσω σαφές. Ε, να μιλήσω και για το θέμα της παρέκκλησης. Δηλαδή, ε, έχει διατυπωθεί το αίτημα η συζήτηση αυτή να διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο. Είπε ένας από τους εμπειρογνώμονες ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, δεν έχει καμία δουλειά να ρυθμίζει τα θέματα των θρησκευτικών κοινοτήτων. Ότι δηλαδή ισχύει η αρχή της επικουρικότητας και θα πρέπει τα θέματα να ρυθμίζονται σε εθνικό ή κοινοτικό ή τοπικό επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνεται μόνο στις χώρες οι οποίες το επιθυμούν. Εάν ο κανονισμός τα απέκλειε όλα αυτά, τότε σίγουρα δεν θα προέβλεπε την ε, συζήτηση του θέματος σε εθνικό επίπεδο μόνο. Ας συζητήσουμε αυτό το οποίο ε, είναι αυτό που λέω εγώ. Αυτό είναι αυτό που λέω εγώ. Ας συζητήσουμε. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τη σήμαση. Η σήμαση του κρέατος είναι πληροφόρηση των καταναλωτών. Δεν έχει καμία σχέση με το ε, ξεδιάλεγμα ή το να δαχτυλοδείξουμε, αν θέλετε, μια συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα. Οι καταναλωτές ζητούν απλώς πληροφορίες και έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν με ποια μέθοδο σφαγιάστηκε το ζώο που καταναλώνουν. Και για ορισμένους καταναλωτές αυτή η πληροφόρηση είναι ζωτική σημασίας. Και αυτή είναι η πρόθεσή μας, δεν είναι πρόθεσή μας να ακτιλοδείξουμε κανέναν. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω και το εξής. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί θα έχουν να κάνουν με τις ε, θρησκευτικές κοινότητες και τις ε, θρησκευτικές σφαγές μόνο. Όμως το σχέδιο κανονισμού δεν είναι αυτή οι μοναδικοί περιορισμοί που υπάρχουν. Θέλουμε να αλλάξουμε τις μεθόδους σφαγιασμού των πουλερικών. Θέλουμε να αλλάξουμε ε, τις μεθόδους σφαγής των ζώων που φέρουν τρίχωμα γούνα. Ένα σωρό περιορισμούς επιβάλλουμε με αυτό το σχέδιο κανονισμού. Και για τους άλλους περιορισμούς γινόμαστε δέκτες παραπώνων και πιέσεων άλλων κλάδων εμπορευόμενων οι οποίοι λένε ότι θα πληγεί η ανταγωνιστικότητά τους, οι οποίοι λένε ότι θα είναι πολύ δυσαρέστη κατάσταση για αυτούς, διότι οι περιορισμοί είναι αυστηρότεροι, οι κανονισμοί είναι αυστηρότεροι και αυτό θα μας καταστήσει λιγότερο ανταγωνιστικούς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι βεβαίως θα πρέπει οι αρχές να είναι ομοιόμορφες και να εφαρμόζονται τόσο στους εγχώριους παραγωγούς όσο και στους εισαγωγείς από τρίτες χώρες και αυτό είναι κάτι που μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Ανεξαρτήτως προέλευσης του κρέατος, είτε προέρχεται από τις τρίτες χώρες είτε από την εσωτερική αγορά, σίγουρα οι προϋποθέσεις θα πρέπει, οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται από όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τη συνεισφορά σας. Ε, ε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ συγκεκριμένα τους τέσσερις εμπειρογνώμονες οι οποίοι πραγματικά έχουν συμβάλει σημαντικά στη σύνταξη του σχεδίου έκθεσης. Πιστέψτε με, θα σεβαστούμε απολύτως τις θρησκευτικέ κοινότητες και τα πιστεύω τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χιράντς Καρσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι οι εμπειρογνώμονες επικεντρώθηκαν ε, ιδιαίτερα στη θρησκευτική διάσταση του θέματος. Θα ήθελα λοιπόν εξ αρχής ε, να πω το εξής. Καλό θα είναι να προβληματιστούμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο, σημείο το, στο επίπεδο το οικονομικό. Η έκθεση αυτή θα επιβαρύνει ε, το θέμα του κόστους και θα επιβαρύνει ένα κλάδο ο οποίος έχει υποφέρει ιδιαίτερος γιατί δεν χρειάζεται να σας θυμίσω πόσα σφαγεία έχουν κλείσει τελευταία. Αυξάνονται τα βάρη των επιχειρήσεων, ζητείτε ε, καινούρια επένδυση από πλευράς επιχειρήσεων, απόκτηση διαφόρων πιστοποιητικών για θέματα καλής διαβίωσης κτλ. Δεν μπορούν, πολλά σφαγεία δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις τόσο επαχθείς απαιτήσει. Ε, μην μιλούμε λοιπόν μόνο για το θρησκευτικό, να επιμείνουμε στο οικονομικό σκέλος του προβλήματος κινήματος, το οποίο είναι σημαντικό και αυτό. Από εκεί και πέρα, από τη στρατηγική σκοπιά, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής ε, των διατάξεων που έχουν να κάνουν με την καλή διαβίωση των ζώων, διότι περιλαμβάνεται ας πούμε και το θέμα της μεταφοράς των ζώων και μιλούμε για πράγματα πολύ περίπλοκα σε κοινοτικό επίπεδο. Ε, όλα αυτά είναι πολύ επαχθή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αφού μας νοιάζει τόσο η καλή διαβίωση των ζώων, τότε γιατί δεν απαιτούμε την ε, να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις ε, τα κρέατα τα οποία ε, τα εισάγουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μήπως εκεί καμπτώμεθα διότι θέλουμε να ενισχύσουμε το διεθνές εμπόριο. Ε, μην είμαστε υποκριτές. Να το παραδεχθούμε. Γιατί δεν αποτούμε τα ίδια από τους υπόλοιπους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν υπάρχουν απαιτήσει τέτοιου είδους από τις τρίτες χώρες. Και άρα ε, καταφέρουμε ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία κρέατος. Ας αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι με αυτές τις καινούργιες διατάξεις θα πλήξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ήδη υποφέρουν τα μάλα. Τέλος, από την ισπανική σκοπιά, σκοπιά του θέματος ε, σας παρακαλώ να προσέχετε τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Ε, άλλο είναι σφαγή και άλλο είναι ε, θυσία στα ισπανικά. Ε, το, η μία έννοια έχει διάφορους συνειρμούς, η άλλη δεν τους έχει. Παρακαλώ λοιπόν να προσέχουμε την γλώσσα μας. Από εκεί και πέρα... Ορισμένα πράγματα δύσκολα εφαρμόζονται στην Ισπανία. Στην Ισπανία το κράτος είναι πολύ αποκεντρωμένο και εμείς αποκεντρώνουμε συνεχώς την κρατική μας εξουσία. Πώς θέλετε να έχουμε εμείς κέντρο αναφοράς. Θέλετε να έχουμε 17 κέντρα αναφοράς σε 17 αυτόνομες κοινότητες για 40 εκατομμύρια συνολικό πληθυσμό. Δεν είναι όλες οι χώρες τόσο κεντρικές χώρες όπως είναι η Πολωνία και θα ήθελα αυτό να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας. Τέλος, από τη θρησκευτική σκοπιά του θέματος να πω τα εξής. γίνεται λόγος για τα δεοντολογικά ζητήματα και ζητήματα ηθικής. Αυτά δεν μας αφορούν ως Επιτροπή Γεωργίας, γιατί ε, ε, ξεφεύγουμε από το πεδίο των αρμόδιοτήτων μας, άρα χάνουμε σε αξιοπιστία. Να αποφύγουμε κίνδυνο ε, θρησκευτικής σύγκρουσης, διαμάχης ή ό,τι άλλου πράγματος. Καλά πάνε τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Βεβαίως θα πούμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με τα διάφορα τελετουργικά ή τυπικά θρησκειών, αλλά από εκεί και πέρα, άπαξ και έχει ε, σφαγιαστεί Άπαξ και έχει σφαγιαστεί και έχει πεθάνει το ζώο, δεν μπορώ να καταλάβω ε, ποια είναι η τυπικα θρησκειων αλλα απο εκει και περα απαξ και εχει σφαγιαστει απαξ και εχει σφαγιαστει και εχει πεθανει το ζωο δεν μπορω να καταλαβω ποια ειναι η διαφορα για το ίδιο. Η διαφορά θα ήταν για τον καταναλωτή που έχει περισσότερες πληροφορίες. Α. Δηλαδή, προκειμένου να καλύψω έναν Ευρωπαίο καταναλωτή θα πρέπει να προσβάλλω ε, και να πλήξω πολύ περισσότερο άλλον καταναλωτή, νομίζω ότι αυτό δεν είναι λογικό. Ε, δηλαδή, δεν θα συμφωνήσω εάν ε, τελικά εκεί καταλήξουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαι σε θέση να συμφωνήσω. Ευχαριστώ. Agnes, please. Ευχαριστώ, η Agnes Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που ε, είναι δυνατόν να έχουμε σήμερα αυτή τη σοβαρή συζήτηση για τον τόσο ευαίσθητο τομέα. Με καθησυχάζει το ότι δεν μιλάμε για το εάν ή όχι θα πρέπει να γίνονται θρησκευτικέ σφαγές, αλλά ε, χαίρομαι που συζητάμε για το πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις Η σα είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς μιλάμε, διότι μιλάμε, πρέπει να μιλάμε για σφαγή των ζώων και όχι για θανάτωση, διότι ε, μιλάμε, τρώμε το κρέας, ε, θα πρέπει λοιπόν να σφάζονται τα ζώα με τρόπο ε, ηθικά σωστό, δεν θα πρέπει όμως ε, να παραμβαίνουμε σε θρησκευτικά ζητήματα. Είμαι ευγνώμων που ο τελευταίος εμπειρογνώμων που μίλησε, δυστυχώς έχω ξεχάσει το όνομά του, Χαίρομαι που είπε ότι ε, χρειάζεται να είμαστε όλοι θετικοί και χαίρομαι επίσης που ανέφερε το θετικό παράδειγμα της Αυστρίας. Όσον αφορά την επισήμανση δεν έχω σοβαρό πρόβλημα. Μου φαίνεται ε, πολύ καλή λύση για να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό και πιστεύω ότι είναι καλό και για τους καταναλωτές γιατί έτσι μπορούν να γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λογική καλή λύση την οποία θα μπορούν να δεχτούν όλοι. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Άγνες. Ο Γκρέφε Τζουμπάριντορφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένας εμπειρογνώμων είπε ότι η σφαγή είναι πάντα απάνθρωπη και πάντα ε, ευάναυση. Απάνθρωποι δεν είναι, το κάνουμε. Είναι κάτι που το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Άλλωστε έτσι έχουμε διασφαλίσει κατά καιρού ε, την ύπαρξή μας. Βάναυσος είναι πάντα ο θάνατος, αλλά το θέμα εδώ δεν είναι το αν είναι απάνθρωπο ή όχι. Το θέμα είναι ε, υπό ποιε συνθήκε γίνεται με τον καλύτερο τρόπο ή με τον χειρότερο τρόπο και πώ μπορούμε να, να ε, λάβουμε υπόψη μα ε, την ευζοία των ζώων. Ε, δεν είμαστε θρησκευτικό κοινοβούλιο, ε, εσείς εκπροσωπείτε την θρησκεία. Ε, έχουμε όμως σήμερα αυτή την ακρόαση Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, κάποιες ε, θέσεις ε, των θρησκευτικών κοινοτήτων, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα και στην συνεδρία των συντονιστών είπα ότι φανατισμός στο θέμα αυτό δεν υπάρχει αποκλειστικά από την πλευρά των θρησκευτικών κοινοτήτων. Συχνά έχω την εντύπωση ότι οι οργανώσεις προστασίας των ζώων συχνά φέρονται με πολύ φανατισμό, με σχεδόν ε, θρησκευτική πεποίθηση. Ε, δεν υπάρχει αιμονή στο κοινοβούλιο μας κατά των θρησκευτικών σφαγών. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Σκεφτόμαστε σοβαρά το θέμα. Δεν έχουμε όμως έμονες ιδέες ως προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ως προς ε, τη θρησκευτική σφαγή λοιπόν. Η αγωνία που περνούν τα ζώα κατά τη σφαγή και στις δύο περιπτώσεις και με και χωρίς αναισθητοποίηση μπορεί να υπάρχει. Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά το γεγονός ότι αυτοί που μιλάνε για θρησκευτική σφαγή παίρνουν πολύ στα σοβαρά την ευζοία των ζώων. Κάτω τη θρησκευτική σφαγή, το ακούσαμε αυτό, ε, απαιτείται εξειδίκευση ε, αυτού που σφάζει ώστε να ε, διασφαλίζεται ότι τα ζώα δεν περνούν ε, από αγωνία και πόνο. είναι ένα θέμα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, στον συγκεκριμένο κανονισμό. Τις συνθήκες δηλαδή όχι μόνο σφαγής, αλλά και τις προηγούμενες, τις συνθήκες που επικρατούν ε, πριν τη σφαγή του ζώου. Κατά τη θρησκευτική σφαγή υπάρχει σεβασμός του ζώου. Ήθελα να το αναφέρω αυτό, διότι Ε, Αλλιώ καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτοί που θέλουν θρησκευτική σφαγή δεν έχουν κανένα σεβασμό για τα ζώα. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Τίθεται το θέμα. Η θρησκευτική σφαγή είναι μεγαλύτερη επιβάρυνση για το ζώο από ότι η σφαγή με, με αναισθητοποίηση. Όπως ε, είπε ο συνάδελφος που ασχολείται με την προστασία των ζώων, ε, μπορεί η αναισθητοποίηση να γίνει μετά ε, την σφαγή και έτσι Φτάνουμε σε ένα, σε συμπέρασμα. Δεν είναι το κόψιμο της καροτίδας ε, το, η ολοκλήρωση της διαδικασίας, είναι η αφέμαξη η κρίσιμη στιγμή. Ε, εγώ έκοψα το δάχτυλό μου. Ε, η πρώτη αντίδραση είναι ότι καταλαβαίνω ότι κάτι έχει γίνει, αλλά τον πόνο τον νιώθω μετά. Δεν είμαι ζώο, άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω αν και τα ζώα περνούν το ίδιο, αλλά εάν υποθέσω ότι Ε, το ζώο νιώθει και αυτό έτσι. Με την ε, κοπή της καροτίδας ε, δεν γνωρίζει ότι έχει σφαχτεί, γνωρίζει ότι κάτι έχει συμβεί. Ίσως λοιπόν η εκ των υστέρων ανιστοποίηση να αποτελεί λύση. Δεν ξέρω αν μπορούν να το δεχτούν αυτό οι θρησκευτικέ κοινότητε, αλλά... Εάν ε, όσοι ε, ενδιαφέρονται για την προστασία των ζώων ε, μπορούν να το δεχτούν αυτό, τότε το βασικό θέμα που μα απασχολεί είναι η αφέμαξη. Εγώ είμαι κυνηγό, σκοτώνω ζώα. Χωρίς αναισθητοποίηση. Δεν πλησιάζω το ζώο να το αναισθητοποιήσω πρώτα. Αναισθητοποίηση γίνεται κατά τη θανάτωση του ζώου. Το αναφέρατε και εσείς αυτό πιθανότατα η θρησκευτική σφαγή να είναι ταυτόχρονη αναισθητοποίηση και θανάτωση. Θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Διότι αλλιώς, Γιώζεφ, ε, θα πρέπει να απαγορεύσουμε και το κυνήγι. Θα πρέπει δηλαδή να σκοτώνουμε τους χείρους με πυροβολισμό, ώστε να φροντίσουμε ότι αναισθητοποιείται το ζώο και με, την, ε, με τον πυροβολισμό και ότι δεν μπορούμε δηλαδή να πυροβολήσουμε αν δεν βεβαιωθούμε ότι το ζώνη ιστοποιείται με, την πρώτη, με τον πρώτο πυροβολισμό. Εάν πούμε ότι δεν δεχόμαστε καμία θανάτωση χωρίς ανιστοποίηση, τότε θα πρέπει να απαγορεύσουμε το κυνήγι. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει πρώτα δηλαδή να, να ε, πυροβολούμε με όπλο ανιστοποίηση. Δεν μπορώ να κρίνω τη θρησκεία σας, αλλά όπως βλέπω εγώ το θέμα, δεν πρόκειται για διάκριση, με κανέναν τρόπο δεν ε, πρόκειται για διάκριση της σχετικής θρησκείας, εάν πρόκειτο για, ε, για διάκριση, τότε αγαπητοί εκπρόσωποι των θρησκευτικών αυτών, τότε θα έπρεπε να έχετε αμφιβολίες για τις θρησκείες σας. Εάν εγώ είμαι πεπισμένος για κάτι, Ε, μπορώ να βάλω ταμπέλα ότι ε, ότι υποστηρίζω αυτά τα πράγματα αλλά έτσι στιγματίζομαι. Ε, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε με τέτοιους όρους. Τουλάχιστον το Κοινοβούλιο ε, δεν θέλει να στιγματίσει, το, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν επιθυμεί να στιγματίσει καμία θρησκεία. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο και ε, θέλουμε να δούμε πόσο ευρύ περιθώριο ευελιξίας έχετε. Και οι θρησκείες εξελίσσονται. Εγώ ως χριστιανός ε, μεγάλωσα. Ε, πριν κάποια χρόνια η ε, χριστιανική θρησκεία έκαιγε γυναίκες επειδή τις θεωρούσε μάγισσες. Ε, έχουμε κινηθεί προς την κατεύθυνση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και έχουμε ξεφύγει από τις ε, θέσεις αυτές. Παρακαλώ λοιπόν και εσάς να το εξετάσετε αυτό. Σας παρακαλώ να δείξετε και εσείς ε, ανεκτικότητα. Εάν όλοι απλά επιμένουμε στις θέσεις μας δεν θα βρεθεί καμία λύση και Εάν η ανιστοποίηση μετά το κόψιμο της καροτίδας αποτελεί λύση για τις θρησκευτικέ κοινότητες, τότε να το εφαρμόσουμε. Και για μένα δεν πρόκειται για θέμα ε, κόστους, δεν μπορούμε να δούμε το θέμα αυτό με οικονομικούς όρους, να δούμε αν στοιχήσει περισσότερο ή λιγότερο. Οι θρησκευτικέ κοινότητε θα πρέπει να δεχτούν τι δαπάνε και εμεί ω ε, Κοσμικό Κοινοβούλιο δεν είμαστε εκπρόσωποι θρησκείας. Δεν είμαι εκπρόσωπος ε, ε, του χριστιανισμού, είμαι βουλευτής. Τυχαίνει να είμαι χριστιανός, ε, αλλά θα μπορούσε ένας βουλευτής τυχαία να είναι Εβραίος ή Μουσουλμάνος. Αλλά πολιτική δεν διαμορφώνουμε υπό το φως των θρησκειών. Δεν ε, θέλουμε να, ε, ε, να καταδικάσουμε καμία θρησκεία. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο για να προχωρήσουμε όλοι μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Κρέφε. Η κυρία Μικέλε Ράμος. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω τη θέση της ομάδας μας ως προς δύο βασικά ζητήματα. σε σχέση με τις τοποθετήσεις των εμπειρογνωμόνων. Πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Η κυρία Έρανς, η κυρία Σρούιμπερ μίλησαν για την θανάτωση και τη σφαγή και την θυσία. Να διευκρινίσουμε λοιπόν το εξής. Μιλούμε για θανάτωση ζώων, για ανθρώπινη κατανάλωση Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ε, σφαγή. Για τα ζώα που θα καταναλωθούν δηλαδή. Και ακριβώς επειδή πρόκειται για ζώα τα οποία ο άνθρωπος θα καταναλώσει, είναι απαραίτητο να έχουμε μία αρμόδια αρχή η οποία θα πιστοποιεί τα κέντρα σφαγής όπου θα θανατωθούν αυτά τα ζώα και η οποία αρχή θα πιστοποιεί ποιος θα υπόκειται σε παρέκκληση. Εξηγούμε, στη χώρα μου, στην Ισπανία, αυτή τη στιγμή, για να γίνουν θρησκευτικές σφαγές ζώων, των οποίων το κρέας προορίζεται για κατανάλωση από ανθρώπους, ε, θρησκευτικές σφαγές λοιπόν, ε, εβραϊκές ή μουσουλμανικές, γίνεται αυτή η θρησκευτική σφαγή σε ξεχωριστά κέντρα που έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή. Γιατί, διότι μιλούμε, επαναλαμβάνω, για κρέας το οποίο προορίζεται ε, για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρόκειται για σφαγή η οποία γίνεται εν είδη θυσίας ή εν πάση περιπτώσει για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Δεν πρόκειται για θυσιαστήρια και θρησκευτικές θυσίες. Μιλούμε για σφαγή ζώων που προορίζονται για κατανάλωση από ανθρώπους να το διευκρινίσουμε. Δεν μιλούμε για θανάτωση αλλά για σφαγή. Και διευκρινίζουμε ότι η σφαγή των ζώων αυτών, ανεξαρτήτως θρησκευτικότητας ή όχι, πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένο σφαγείο από την αρμόδια αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριο Στόλ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση. Απλώς θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτά που πάνε οι, προς, οι προλαλήσαντες, όπως είπε και ο Γκρέφ, ε, για το κυνήγι, ας πούμε. Εντάξει, βέβαια το κυνήγι δεν είναι το ίδιο πράγμα με τα ζώα που πηγαίνουν ε, σε εγκαταστάσεις ε, που έχουν ελεχθεί. Μιλάμε για ένα σύστημα ε, σφαγής, για ένα σφαγείο υπάρχει έλεγχος από τις διάφορες αρμόδιες αρχές ε, και από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των κρατών και δεν καταλαβαίνω λοιπόν ε, γιατί υπάρχει πρόβλημα με όλο αυτό. Εντάξει, μετά να κάνουμε όλες τις αναλύσεις που θέλετε να κάνουμε, αλλά αν δεν δεχόμαστε αυτό που γίνεται ε, στα σφαγεία που επισήμως ελέγχονται, εγώ είμαι πρόεδρος σφαγείων και ξέρω τι γίνεται. Έχουμε συγκεκριμένες μεθόδους ώστε να υποφέρει όσο το δυνατόν γίνεται, όσο το δυνατόν λιγότερο το ζώο. Ούτως ή άλλω όσοι γνωρίζουν από σφαγεία θα ξέρουν ότι δεν τρώγεται το κρέα όταν υποφέρουν τα ζώα. Αν ε, σπάσουν τα αγκία, αν υπάρχει κακή μεταχείριση του ζώου ή αν μεταφέρεται με κακές συνθήκες το ζώο στον τόπο σφαγή. Ε, Εκείνο που καταναλώνει το κρέα, που το αγοράζει, είναι αυτό που υποφέρει και το γνωρίζουμε καλά. Οπότε έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε σε επίπεδο σφαγίου, ώστε τα ζώα ε, δεν θα αναφέρομαι. Εντάξει, δεν, δεν, δεν, υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι έχουμε λάβει ούτως ή άλλως όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σφαγιάζονται σωστά ε, και έχουμε σεβαστεί τις αξίες και τις παραδόσεις που είναι ε, πάνω στις οποίες βασίζεται η κοινότητά μας. Ε, γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει. Εκεί είναι που πρέπει να κάνουμε, να, να, δούμε, να, δούμε τα πράγματα προσεκτικά. Αν ε, δεν είναι σωστές οι μέθοδοι ελέγχου από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, θα έχουμε εμείς πάλι πρόβλημα και στην Ήπεθρο και στο δάσος και παντού. Αυτό θέλουμε να γίνει, να σεβόμαστε τις παραδόσεις και τις αξίες μας με σφαγεία, τα οποία έχουν το σωστό εξοπλισμό έχουν πάρα πολλά ε, χρήματα δαπανηθεί ώστε τα πράγματα να γίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό ήθελα να πω σε σχέση με τα σφαγεία. Λοιπόν, πρέπει να αποκλείσουμε. Πραγματικά έχω βαρεθεί να ακούσω, να ακούω από πού έρχονται οι κριτικές, ε, οι περισσότερες κριτικές που έρχονται κατά των ε, σφαγίων είναι από τους από τους ε, χορτοφάγους ε, οι οποίοι δεν τρώνε κρέας ε, και δεν θα πω τίποτε παραπάνω για να μην ξεφύγω από τα, ξεφύγω από τα όρια της ευγένειας. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το σύστημα με τους επιστήμονες, με τους κτηνιάτρους. Βεβαίως επιδέχεται βελτιώσεων το όλο σύστημα. Ευχαρίστως να το ακούσω. Ακόμη στα σφαγεία, βεβαίως. Απλώς θέλω να πω να μην φτάσουμε και στα άκρα, να αποφύγουμε τα άκρα. Αυτά ήθελα εγώ να προσθέσω ως προς το θέμα αυτό, να μην έχουμε ένα σύστημα θρησκειών, να μην έχουμε ένα σύστημα ακραίο τέλο πάντων, δουλεύουν καλά τα σφαγεία, υπάρχει επιθεώρηση, υπάρχει επιστημονική παρακολούθηση, υπάρχει κτηνιατρική παρακολούθηση, να συνεχίσουμε έτσι και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα ε, όσο μπορούμε. Δεν χρειαζόμαστε 25 παραπάνω νομοθεσίες για να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντζαρέλο και μετά ο κύριος Αντός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα αυτή να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες για να έχουμε καλύτερη κατανόηση του λεπτού αυτού ζητήματος. Όσον αφορά την ευζοία των ζώων, έχουν γίνει πολλά στον τομέα της εκτροφής και της μεταφοράς. Τώρα προχωράμε πιο πέρα. Ασχολούμαστε με το στάδιο της φαγής. Για να διασφαλίσουμε την ύπαρξη μη βάναυσων διαδικασιών θανάτωσης πολιτισμένων μεθόδων. Επί Κεντρωνόμαστε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα μόλις ταλαιπωρίες κατά τη στιγμή της φαγής τους. Και το θέμα είναι αν παραβιάζουμε βασικές αρχές. Ε, μιλάμε για βασικές αρχές ε, θρησκευτικών πρακτικών, ε, Ισλαμικών και Εβραϊκών. Στην Ιταλία έχω διαβάσει στον τύπο για το θέμα αυτό. Ε, είναι ένα θέμα που τονίστηκε κατά την ε, ε, Ισραηλινή προεκλογική εκστρατεία. Θεωρήθηκε σκάνδαλο ότι κάποιος πολιτικός ηγέτης δεν σεβάστηκε τις αρχές για το φαγητό κόσερ. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις θρησκευτικές πεπιθήσεις και θρησκευτικές διαδικασίες των ανθρώπων. Δεν είναι δευτερεύοντα τα ζητήματα που συζητάμε. Είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Όταν μιλάμε για θρησκευτικέ ε, σφαγές, ε, εάν φροντίσουμε ε, να τηρούνται τα πρότυπά μας, εντάξει θα πρέπει όμως να είμαστε συνεπείς. Δεν μπορούμε να επιμένουμε στην αναισθητοποίηση και στην σφαγή ε, όταν είναι όρθιο το ζώο. Πρόκειται για βασικές ε, αρχές και έχουν ε, διαμορφωθεί για θρησκευτικούς λόγους με συγκεκριμένο τρόπο η διαδικασία σφαγής. Δεν αρκεί να πούμε ότι α, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ο κύριος Ντόλ νομίζω το είπε αυτό έτσι. ουσιαστικά θα ενθαρρύνουμε τις παράνομες ε, σφαγές ε, και ε, σφαγές στα κρυφά, στα σφαγεία. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση, θα πρέπει και από τις δύο πλευρές να υπάρχει κατανόηση. Δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την παράνομη σφαγή ζώων. Να σκοτώνει κανείς ζώα στο μπάνιο του ή στο δάσος. Θα πρέπει η όλη συζήτηση να στηριχτεί στην αμοιβαία, στον αμοιβαίο σεβασμό. Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα και στις εισαγωγές. Θα πρέπει δηλαδή να ζητάμε από τρίτες χώρες να σεβαστούν τα ίδια πρότυπα. Θέλουμε αμοιβαιότητα. Εάν ε, όμως τελικά καταστεί, ε, ε, αδύνατη η εισαγωγή τροφίμων κόσερ ή χαλάλ, Αυτό θα είναι πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για απαιτήσει προ τρίτε χώρε. Θα πρέπει πράγματι να υπάρχει αμοιβαιότητα. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για λίγα δευτερόλεπτα όπου είναι πιθανό να ταλαιπωρείται το ζώο. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό όμως επιστημονικά. Ε, διατηρήσουμε λοιπόν την ψυχραιμία μας, ας αποφύγουμε ε, να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ε, σκοτώνει, ε, να σφάζει με παράνομους τρόπους τα ζώα. Επίσης όσον αφορά την επισήμανση. Οι καταναλωτές σε διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων θέλουν να αγοράζουν από σούπερ μάρκετ όπου είναι βέβαιοι ότι το προϊόν προέρχεται από σφαγεία που σφάζουν με τον τρόπο που το επιθυμούν. Θα πρέπει δηλαδή να ε, διασφαλίσουμε τις εγγύησεις αυτές. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε ε, να ε, καταδεικνύουμε με μετροπιαστικό τρόπο τις θρησκευτικέ κοινότητες. Είμαι σκιώδης στο θέμα αυτό. Έχω ασχοληθεί με κάποια επίμαχα σημεία στο θέμα της προστασίας των ζώων. Με βάση τη δική μου εμπειρία Ε, θα έλεγα ότι πρέπει να μην έχουμε έμονες ιδέες κατά τις εφαρμογές. Ε, θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και, ε, διότι αν βιαστούμε δεν θα βοηθήσει αυτό τις θρησκευτικέ κοινότητες. Ευχαριστώ κύριο Καπλασάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε πρόβλημα είναι πολυδιάστατο και οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται μετά από ενδελεχή ανάλυση όλων των πτυχών ενός ζητήματος. Το θέμα που μας απασχολεί έχει θρησκευτική διάσταση, αλλά έχει και οικονομική διάσταση και έχει και άλλες διαστάσεις πολύ σημαντικές. Ε, δεν θέλω να αναφερθώ σε όλες αυτές. Το μόνο που θέλω να πω σήμερα είναι το εξής. Δεν λέω ότι το δικό μου παράδειγμα πολιτισμού είναι ανώτερο των άλλων. Λέω όμως ότι έχουμε κοινότητα ε, εθνών και κρατών όπου υπάρχει θρησκευτική ανέξη θρησκεία, όπου υπάρχει σεβασμός των μικρών κοινοτήτων από τις μεγαλύτερες κοινότητες. Εδώ μιλούμε για τη θέση μας ως προς την οδύνη των ζώων. Αυτό είναι αυτό που συζητούμε την οδύνη των ζώων. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως πώς ακριβώς θανατώνεται ένα ζώο. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να θανατώνεται με τρόπο ο οποίος θα ελεγχιστοποιεί την οδύνη την οποία βιώνει. Ανεξαρτήτως του αν η μέθοδος σφαγής ε, πόρο απέχει ή ε, πολύ προσεγγίζει τις απαιτήσει ε, του θρησκευτικού τυπικού. Θα επανέλθω όμως αυτά. Ε, μιλούμε ε, για θέματα επίσης οικονομικά, για θέματα οικονομικής ασφάλειας, για την άνοδο του κόστους, για την ε, άνοδο της ακρίβειας, για την ασφάλεια των εργαζομένων επίσης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πραγματικά στοιχεία. Η θρησκευτική σφαγή βάσει των ευρω... ευρωαϊκών ή μουσουλμανικών προτύπων προκαλεί την περισσότερη οδύνη ή όχι. Αν προκαλεί ε, την ίδια οδύνη ε, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα από τη στιγμή που γίνονται σεβαστοί οι κανόνες υγιεινής κτλ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιβάλλουμε περιστροφές εναλλαγές μόνο επί τη βάση θρησκευτικών αιτημάτων. Ιδελώς θα έχουμε διακρίσεις απαράδεκτες. Ζητώ λοιπόν περισσότερες διευκρινήσεις. Ερωτώ, ε, κάποια συστήματα, κάποιες μέθοδοι σφαγής προκαλούν περισσότερο ή λιγότερο. Υπό αυτό το πρίσμα να εξετάσουμε την κατάσταση. Ο πρόεδρος, να ε, πω δύο λόγια κι εγώ παρακαλώ και να δώσω ξανά το λόγο στους εμπειρογνώμονες για δύο-τρία λεπτά. Λοιπόν, εδώ έχουμε συγκεντρωθεί για να συζητήσουμε ε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μειωθεί η οδύνη των ζώων τα οποία προορίζονται για σφαγή. Αναμφισβήτητα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και σε διάφορα μέρη του κόσμου σφαγιάζονται ζώα με διαφορετικούς τρόπους με διαφορετικές θρησκευτικέ φαγές με αναισθητοποίηση πριν ή μετά τη σφαγή. Κάποια από τα ζώα αυτά χαρακτηρίζονται ως ζώα κοσέρ, άρα μπορούν να καταναλωθούν με βάση συγκεκριμένες θρησκευτικέ επιταγές, κάποια άλλα όχι. Ε, κάνουμε όμως εισαγωγές. Ε, για παράδειγμα, η Μαλαισία δέχεται κρέας ε, εισαγόμενο από Αυστραλία από άλλες χώρες και το δέχεται ως κοσέρ. Προσπαθούμε λοιπόν εδώ να ε, κάνουμε το σύστημα το ευρωπαϊκό πιο ομοιόμορφο, να το εναρμονίσουμε αν θέλετε κάπως. Αναζητούμε μια συμβιβατιστική λύση, δεν επιδιώκουμε να δώσουμε ένα τέλος την θρησκευτική σφαγή, να την εξαλείψουμε από προσώπου Προσπαθούμε να ε, συμβιβαστούμε στην εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων αναισθητοποίηση για να μειώσουμε στο ελάχιστο την οδύνη των ζώων. Ερωτώ λοιπόν γιατί αυτό είναι εφικτό ε, σε κάποιες χώρες και σε κάποιες άλλες όχι. Είναι θέμα ε, θρησκευτικού νόμου, ερωτώ τους πάντες, είναι δυνατό κάτι τέτοιο και αναφερθήκατε και στο άρθρο 4 του σχεδίου κανονισμού. Κοιτάξτε, εμείς στην Επιτροπή ε, Γεωργίας μιλούμε για υψηλά πρότυπα παραγωγής και προστασίας. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο ότι τα δικά μας πρότυπα είναι υψηλότερα των άλλων χωρών, ειδικότερα ως προς τις εισαγωγές. Οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ε, την ύπαρξη, τη θέσπιση αν θέλετε κανόνων που εξασφαλίζουν ότι έχουμε πραγματικά υψηλά πρότυπα τα σφαγεία μας. Αλλιώς ε, δεν ε, έχουμε κανένα επιχείρημα ε, για να αντιπαραθέσουμε στις τρίτες χώρες. Και τρίτη μου παρατήρηση, γιατί αρκετοί από εσά είστε τόσο εναντίον της σήμανσης. Τι διαφορά σας κάνει, δεν σας ε, επιβάλλουμε καμία διάκριση, δεν σας δαχτυλοδείχνουμε. Αν εσείς πουλάτε το κρέας ως κοσέρ, κρέας που μπορεί να καταναλωθεί δηλαδή από την εβραϊκή κοινότητα, τότε θα πρέπει να φαίνεται αυτό στη σήμανση, να το ξέρει ο κόσμος για να μπορέσει να το αγοράσει όποιος θέλει. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει η αντίθεσή σας στη σήμαση, στην υποχρέωση σήμασης και ελπίζω να μην είναι οικονομικού χαρακτήρα η διαφωνία σας. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα το απόγευμα. Προσπαθούμε, επαναλαμβάνω, να επιδιώξουμε μια συμβιβαστική λύση η οποία θα είναι αποδεκτή για όλους μας ώστε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας. Να ξεκινήσω με τον πρώτο εμπειρογνώμονα για την ε, απάντησή του. Κύριε Νόγκα, τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Okay. Um, if possible, I will speak in ε, θα προτιμήσω να μιλήσω Ιταλικά. Ευχαριστώ. Την ερώτηση για την ανιστοποίηση μετά το κόψιμο της καροτίδας ε, θα το αφήσω στους εκπρόσωπους της συσκευτικής κοινότητας, αλλά ως προς την επισήμανση προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα θα είναι επιρροή στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στην κανονική σφαγή και τη θρησκευτική σφαγή. Οι περισσότεροι, ακόμα και φίλοι μου κτηνίατροι από το Πανεπιστήμιο, δεν γνωρίζουν τη διαφορά. Νομίζουν ότι η θρησκευτική σφαγή είναι βάρβαρη. Πιστεύουν ότι το ζώο υποφέρει. ενώ πιστεύουν ότι με την αναισθητοποίηση δεν υποφέρει καθόλου το ζώο. Δεν γνωρίζουν λοιπόν τη διαφορά. Δεν είναι αλήθεια αυτά. Εγώ ως κτηνίατρος θα έλεγα ότι υπάρχει διαφορά. Ο Ιταλός βουλευτής το είπε. Μιλάμε για λίγα δευτερόλεπτα διαφοράς. Προσπαθώ δηλαδή να πω ότι προτού προχωρήσουμε στην επισήμανση θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ώστε να γνωρίζει ποια είναι η διαφορά, στην οποία περίπτωση δεν θα αποτελέσει πρόβλημα η επισήμανση. Όσο όμως ο περισσότερος κόσμος αγνοεί την είναι η θρησκευτική σφαγή, ε, η επισήμανση μπορεί να οδηγήσει σε στιγματισμό και σε διάκριση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φίσον. Εκτός μικροφώνου μιλητής. Λοιπόν, όσον αφορά τη σήμανση Κοιτάξτε, η κατανάλωση του κρέατος κόσερ προέρχεται από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Μιλάμε για σήμανση κρέατος που προορίζεται για το ευρύ κοινό. Εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, στη Γαλλία σε σχέση με ακραίες οργανώσεις προστασίας ζώων. Δεν μιλάω για συναδέλφους με τους οποίους έχουμε πολύ καλές σχέσεις ε, και με τους οποίους προσπαθούμε να βρούμε από κοινού λύσεις, αλλά Υπάρχουν πολύ ακραίες οργανώσεις προστασίας των ζώων που θα εκμεταλλευτούν αυτές τις διατάξεις για εκστρατείες, για να στιγματίσουν, για να καταδείξουν την εβραϊκή κοινότητα και θα πει ωραία ε, κοινότητα εβραϊκή, κοινότητα ε, μουσουλμανική, τι κακοί άνθρωποι σφάζουν τα ζώα χωρίς ε, αναισθητοποίηση. Κάποιος ανέφερε το θέμα της αναστητοποίησης και ανέφερε κατά πόσο είναι επιπλέον ε, προστασία των ζώων. Για μερικούς αυτό είναι προφανές, για άλλους όμως όχι και σας το λέω αυτό γιατί υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία. Δεν είναι σαφές αυτό. Ε, υπάρχουν εμπειρίες ε, υπέρ, υπάρχουν εμπειρίες κατά, υπάρχουν και επιστημονικά στοιχεία υπέρ και κατά τι είναι το καλύτερο για την ευημερία των ζώων. Είναι η κοπή, η τομή της καροτίδας, είναι η εκ των προτέρων αισθητοποίηση. Ούτως ή άλλως ε, η αναισθητοποίηση πριν ή μετά τη σφαγή δεν μας είναι αποδεκτή, δεν τη δεχόμαστε γιατί υπάρχουν κανόνες θρησκευτικοί Σα το εξήγησα για την αναισθητοποίηση και πριν και μετά. Υπάρχει το θέμα της αφέμαξης που πρέπει να είναι πλήρης. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επιβάλλει αυτούς τους κανόνες και της σήμανσης, ε, θα τίθεται ένα αμφιβόλο η θρησκευτική σφαγή. Δεν ε, είπα ότι είναι εναντίον της μίας ή της άλλης θρησκείας και είπατε κι εσείς ότι είναι θέμα μόνο προστασίας των ζώων, αλλά πραγματικά είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να πνίγουμε, για να το πω έτσι, το, τη θρησκευτική σφαγή, σαν να προσπαθούμε να την ε, κουκουλώσουμε. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι αυτή η πρόθεση. Καταλαβαίνω ότι η πρόθεση δική σας ε, είναι η προστασία των ζώων, αλλά είναι ουσιαστικά απαγόρευση το, της ε, κατανάλωσης ε, του κρέατος της εβραϊκής και της μουσουλμανικής κοινότητας. Μην μας επιβάλλετε κανόνες που δεν θα μπορέσουμε να ε, σεβαστούμε. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει το θέμα της προστασίας των ζώων, αυτό το δεχόμαστε απόλυτα, αλλά ως προς τις λεπτομέρειες του πράγματος είμαστε μάλλον απογοητευμένοι ε, από την πορεία της συζήτησης. Πρόεδρος, κοιτάξτε, η ερώτηση που δεν απαντάτε είναι γιατί σε μερικά κράτη-μέλη γίνεται ε, σφαγή των ζώων με εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων υπό το θρησκευτικό νόμο όμως. Είτε είναι κόσερ, είτε είναι χαλάλ, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια διαδικασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η απάντηση που δεν μου δίνεται. Μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Κοιτάξτε, η αναισθητοποίηση, θα το επαναλάβω. Η αναισθητοποίηση πριν από τη σφαγή ή αμέσως μετά τη σφαγή ε, κάνει το κρέας μη, όχι, ε, όχι κόσερ και δεν μπορούμε εμεί πλέον να καταναλώνουμε αυτό το κρέας που δεν είναι κόσερ. Αυτό σας εξηγώ. Πρόεδρος, μάλιστα. Οπότε δεν ε, χρησιμοποιείτε, δεν καταναλώνετε κρέας από τι άλλε χώρε που ακολουθούν αυτό το σύστημα. Αμφιβάλλω, αλλά αυτό μας λέτε ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που θέσατε και στα άλλα ερωτήματα που ετέθησαν όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία της θρησκευτική φαγής είναι κάτι το οποίο θέσατε πολύ πρόσφατα. Εγώ αμφισβητώ τα αριθμητικά αυτά στοιχεία. Εντάξει, δεν θα μπούμε τώρα σε μία μάχη αριθμητικών στοιχείων ε, αλλά η Γενική Διεύθυνση ε, Τροφίμων της Γαλλίας ε, έχει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Στη Γαλλία η κατανάλωση κρέατος ε, βοδινού είναι το 168% του συνολικού κρέατος, δηλαδή δύο στα τρία σφάγια ε, είναι εισαγόμενα στη Γαλλία. Όσον αφορά το βόλιο κρέας, ε, βρισκόμαστε σε μια ισοδυναμία σχεδόν. Έχουμε 11% 13% ε, είναι οι ε, σφαγές. Υπάρχει δηλαδή μία ισορροπία στη Γαλλία. Δεν ε, υπάρχει λόγος να αναφέρουμε απλώς αριθμητικά στοιχεία χωρίς να λέμε τι σχέση έχουν με το ευρύτερο πλαίσιο. Και σας μιλάω τώρα για στοιχεία του γαλλικού κράτους. Τώρα για την ερώτηση που κάνατε σε σχέση με τη διαφορά μεταξύ των χωρών. Κοιτάξτε, Υπάρχουν ε, θρησκευτικές αρχές, υπάρχει το Κοράνι. Πώς να σας το πω τώρα. Ε, δεν... Ε, η, η, η θρησκεία είναι αυτή που επιβάλλει αυτούς τους κανόνες. μπορώ να σας εξηγήσω για ποιο λόγο υποφέρει όχι το ζώο λιγότερο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι είναι θεματοφύλακας του δικαιώματος τη ανεξιθρησκείας και εμεί είμαστε πεπισμένοι Ευρωπαίοι είμαστε τμήμα του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αναπόσπαστο τμήμα, Τις 29 Ιανουαρίου ετέθη ένα ερώτημα από έναν βουλευτή. Δεν είναι ισχυρισμοί. Η κυρία Μουσκαρντίνη έκανε αυτό το ερώτημα. έχει αναφερθεί ότι είναι βάναυσος ο τρόπος που θανατώνονται τα ζώα αυτά. Ότι είναι μια βάρβαρη πρακτική ανέφερε. Κοιτάξτε, είναι πράγματα που έχει πει η βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ ε, πρέπει να πω ότι υπάρχει αυτό το κλίμα. Δεν ε, το βγάζω από το μυαλό μου. Έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα και πρέπει να, να είμαστε λίγο προσεκτικοί ως προς αυτό. Εμείς μόνο για το άρθρο 4 μιλάμε. Τα υπόλοιπα θέματα για μας ε, έχουν προοδεύσει αρκετά, αλλά το άρθρο 4 δημιουργεί πρόβλημα στη θρησκευτική σφαγή. Μιλάμε για την Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που πρέπει να ε, δημιουργούν τους ε, κανόνες και δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε σε χώρες εκτός Ευρώπης για να δούμε τι κανόνες θα ισχύσουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Ευχαριστώ. να σας πω. Question from one member of this Να σας πω ότι μία βουλευτής έκανε μία συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι απηχεί τις απόψεις ε, του συνόλου του σώματος. Δεν έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε θρησκευτική βεντέτα. Είμαστε εδώ για να βρούμε μια κάποια λύση Κάποιες χώρες χρησιμοποιούν την εκ των υστέρων αναισθητοποίηση. Γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς. Δεν έχετε κατεφέρει να με πείσετε ακόμα. Παρακαλώ, τελευταίος εμπειρογνώμονας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να συνεχίσουμε αυτή την ε, στέρφα συζήτηση. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Θα ήθελα να πω μόνο το εξής. Δεν τοποθετούμε για θρησκευτικά ζητήματα. Λέω όμως το εξής. Λέτε ότι το κρέας δεν είναι πια κοσέρ όταν γίνεται η ανισοτοποίηση μετά τη σφαγή. Οι ραβίνοι όμως της Αυστραλίας λένε ότι είναι κοσέρ. Και σε διάφορα άλλα ε, μέρη στην Αγγλία Υπάρχει επίσημη έκθεση που λέει ότι η αναισθητοποίηση μετά τη σφαγή είναι κοσέρ, μπορεί να καταπολεμηθεί. Λοιπόν, θα ήθελα κάποιος να μου απαντήσει. Είναι σημαντικό αυτό. Η εκ των υστέρων αναισθητοποίηση είναι λύση. Λύση και για τη μείωση της οδύνης των ζώων. Δεν είναι μόνο θρησκευτικό το πρόβλημα, είναι και επιστημονικό, είναι κτηνιατρικό θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαιτέρως. Λέω λοιπόν ότι δεν γίνεται πλέον συζήτηση για τη σήμαση, διότι εάν κάνουμε αναισθητοποίηση μετά τη σφαγή θα ισχύσει για όλα τα ζώα και θα πούμε στο καταναλωτή ότι τα ζώα ανεσυντοποιούνται τη στιγμή της σφαγής. Άρα με ένα σπάρο δυο τριγώνια πετυχαίνουμε. Είναι συμβαστική λύση αυτή, καλή. Λύνονται προβλήματα. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας. Μπορεί να θεωρηθεί το κρέας κοσέρ ακόμα και με την ε, μετά τη σφαγή. Από εκεί και πέρα, εξαιρετικά σημαντικό είναι να έχουμε σαφείς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κάποιες ε, χώρες ήδη εφαρμόζουν αυτά τα πρότυπα. Δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα αυτό για μας από τη στιγμή που υιοθετούμε μια ξεκάθαρη γραμμή στάσης. Εγώ πιστεύω ότι η αναισθητοποίηση μετά τη σφαγή είναι η βέλτιστη συμβαστική λύση για όλα τα θέματα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή και σας ευχαριστώ όλους όσοι ήρθατε να παρουσιάσετε τα επιχείρηματά σας. Ο εισηγητής θα συντάξει το, τη, τη τελική πρόταση έκθεσης, την οποία και θα εξετάσουμε. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 19 Φεβρουαρίου, στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Και θα ψηφίσουμε στις 16 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας. Και θα περιμένουμε με αγωνία την έκθεση του Γιάννους. Γιάννους, μήπως θα ήθελες να κάνεις κάποια τελευταία παρατήρηση. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θέλω να καταστήσω σαφές για άλλη μια φορά το εξής θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόταση δική μας είναι μία βούληση, είναι η βούληση για την επίτευξη συμβαστικής λύσης. Αν δείτε την πρόταση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής θα δείτε ότι η πρόταση αυτή πηγαίνει πολύ πιο πέρα και απαγορεύει στη θέμελα την θρησκευτική σφαγή. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο και ε, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να επιτύχουμε συμβαστική λύση και θα πρέπει ως προς το τι θα προβλέπετε ε, ως παρέκκληση και τι όχι να εξετάσουμε το γεγονός ότι ορισμένες χώρες έχουν θεσπίσει άλλους κανόνες για τη θρησκευτική σφαγή. Και εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας Θεμάτων Αγροτικών Σφαϊκού Κοινοβουλίου ε, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να οπισθοχωρούμε ούτε να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε τις χώρες που θέλουν να επιβάλλουν πιο αυστηρούς περιορισμούς. Τώρα, ουδής αμφισβητεί τη θρησκευτική ελευθερία. Ουδής αμφισβητεί το ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία εντάσσονται στην εθνική αρμοδιότητα, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν μπορεί να παρέμβει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πεδίο αρμοδιότητας των εθνικών αρχών. Θέλουμε λοιπόν να παραμείνει το άρθρο 4 ως έχει, το πνεύμα του δηλαδή, το περιεχόμενό του να ε, παραμείνει ως έχει. Άλλωστε είναι ένα άρθρο το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι δύσκολο να αλλάξει κάτι σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ τον Γιάννου, σας ευχαριστώ όλους θερμά ε, για την συνεισφορά σας. Θα ε, συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε την έκθεση εν ευθέτω χρόνο. Προχωρούμε λοιπόν. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, παρακαλώ αν δεν ενδιαφέρεστε να αποχωρήσετε από την αίθουσα ησύχως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εξέταση του σημείου 5 της ημερήσιας διάταξης. Προστασία ζωών που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Ο υποφαινόμενος είναι η εισηγητής για την Επιτροπή Θεμάτων Γεωργίας. Έχουμε γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, Έρευνας και ε, Έχουμε προσκαλέσει λοιπόν τρεις εμπειρογνώμονες για τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων, οι οποίοι και θα σχολιάσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ε, τους ελέγχους και τις ε, δοκιμές σε ζώα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πάτρικ, ο οποίος δούλεψε τόσο πολύ και ο οποίος έχει συγκροτήσει μια πολύ περίπλοκη έκθεση. Έχουμε υποβάλει πάρα πολλές τροπολογίες στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων μας σήμερα το απόγευμα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έπρεπε να βρεθώ ενώπιον ενός τόσο μεγάλου ηθικού διλήμματος. Θέλω να μειώσω όσο το δυνατόν περισσότερο τις δοκιμές σε ζώα. Θέλω όμως να είμαι βέβαιος ότι θα γίνονται όλο και περισσότερες δοκιμές των φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους στο μέλλον ώστε να είναι ασφαλή. Είναι δύσκολο, λοιπόν, είναι δύσκολο το τέριασμα αυτό των δύο. Θα ακούσουμε από εμπειρογνώμονες. Καταρχάς τον δόκτωρα Μάρκ Μάτφιντ, Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βιοιατρικής Έρευνας. Κύριε Μάτφιτ, σας, δίνω αυτή αμέσως το λόγο. Έχετε 10 λεπτά, παρακαλώ να μην τα ξεπεράσετε. Ευχαριστώ. Mr. Chairman, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων που μου δίδεται η δυνατότητα να μιλήσω στην Επιτροπή σας σήμερα. Είμαι επιστήμονας που εργάζεται στον τομέα των ερευνών ε, για τον καρκίνο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα όμως εκπροσωπώ ε, τους ακαδημαϊκούς επιστήμονες που εργάζονται στα ε, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μας είναι θεμελιώδης έρευνα, πώς λειτουργεί το σώμα μας και τι πάει στραβά όταν ε, αρρωσταίνουμε. Η ε, βασική έρευνα δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξη νέων ε, φαρμάκων ή θεραπείων, αλλά θα ήταν αδύνατον για τις φαρμακευτικές εταιρείες μας να αναπτύξουν νέες θεραπείες και νέα φάρμακα χωρίς τις γνώσεις που προέρχονται από τη θεμελιώδη έρευνα. Ίσως μερικές φορές ο κόσμος παραβλέπει πόσο σημαντική είναι η ακαδημαϊκή έρευνα Επιτρέψτε μου λοιπόν να τονίσω ότι οι ακαδημαϊκοί ερευνητές ανακάλυψαν την πενικυλίνη, ε, ανέπτυξαν ε, τα, τους πρώτους υπολογιστές και το διαδίκτυο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Ε, ακαδημαϊκοί ερευνητές εξερεύνησαν το γονιδίωμα, ανακάλυψαν την αιτία του AIDS και του καρκίνου στον δικό μου τομέα. Το θέμα με τέτοιου τύπου έρευνα είναι ότι ε, προχωράμε στο άγνωστο. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μέχρι να το βρούμε. Ε, γι' αυτό ακριβώ η ελευθερία επιστημονική έρευνα είναι τόσο σημαντική. Κανεί δεν ξέρει ε, ποια θα είναι τα σημαντικά βήματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό οι ερευνητέ αυτοί να έχουν την ελευθερία να ακολουθήσουν την πορεία που θεωρούν ότι είναι σημαντική. Βέβαια σε μια δίκαιη κοινωνία θα πρέπει να υπάρχουν όρια στην ε, ελευθερία αυτή διότι θα πρέπει να είναι ηθική και νόμιμη η έρευνα αυτή και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε την πρόταση οδηγίας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία της πρότασης τα οποία θεωρούν πολύ καλά οι ακαδημαϊκοί ε, ερευνητέ. Ε, συμμετείχαν σε διαβούλευση κατά την ε, προκατακτική φάση. Είναι όμως υπερβολικά γραφειοκρατικό αυτό που προτείνεται. και επιβάλλεται ε, αδικαιολόγητο γραφειοκρατικό άχθος ε, στους ε, ερευνητές. Τα κράτη-μέλη επενδύουν σημαντικά χρηματικά ποσά στην ακαδημαϊκή έρευνα και είναι προφανές ότι θέλουμε οι επιστήμονες να ξοδεύουν το χρόνο τους κάνοντας επιστημονικά πειράματα, όχι συμπληρώνοντας έντυπα. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν κάποια σημεία όπου η πρόταση ε, αντιπροσωπεύει η παρεξήγηση της διαδικασίας ε, της ε, έρευνας και έτσι προτείνει κάποια μέτρα τα οποία θα βλάψουν σημαντικά κάποιους τομείς σημαντικών ερευνών που διεξάγονται στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα οι λέξεις ε, αυτές οι τελευταίες ε, έχουν να κάνουν με το πώς ε, λειτουργεί ο εγκέφαλος. Η κοινωνία στην Ευρώπη γερνάει. Όσο μακραίνει η ζωή μας, τόσο περισσότερες ασθένειες έχουμε όπως επιληψία, Alzheimer, εγκεφαλικά, σχιζοφρενία και άλλες ασθένειες του εγκεφάλου. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αποτελεσματικές θεραπείες θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς εργάζεται ο εγκέφαλος. Αυτό συχνά σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε ε, μη ε, ανθρώπινα πυθικοειδή. Και ο άνθρωπο είναι πυθικοειδέ. Ε, υπάρχουν λοιπόν σημαντικέ ομοιότητε ανάμεσα στου εγκεφάλου μα και του εγκεφάλου των ζώων αυτών. Μιλάμε για έρευνε οι οποίε δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε κανένα άλλο ζώο λόγω των ανατομικών και φυσιολογικών διαφορών στου εγκεφάλου. Αν χρησιμοποιήσει κανεί οποιοδήποτε άλλο ζωικό είδο, τα αποτελέσματα δεν θα είχαν κανένα νόημα. Η πρόταση αυτή λοιπόν ε, προτείνει δύο ε, περιορισμούς ε, που δεν είναι πολύ σοφοί. Καταρχήν στο άρθρο 8 προτείνει να περιοριστεί ο αριθμός επιθυκοειδών στις έρευνες αποκλειστικά στις ασθένειες που απειλούν την ζωή ανθρώπων ή την επιμερία τους. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται οποιαδήποτε έρευνα έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και αυτή η έρευνα είναι ζωτική σημασία αν θέλουμε στο μέλλον να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα σε φυσιολογική λειτουργία εγκεφάλου και μη φυσιολογική λειτουργία εγκεφάλου, σε περίπτωση δηλαδή ασθένεια του εγκεφάλου. Το δεύτερο θέμα, κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με την εκτροφή. Ε, των πυθικοειδών. Όλα τα πυθικοειδή που χρησιμοποιούνται ε, στις έρευνες στην Ευρώπη εκτρέφονται ε, ειδικά για τις έρευνες αυτές. Ε, στο άρθρο 10 της προτινόμενης οδηγίας προτείνεται να να περιοριστούν οι έρευνες στα ζώα που εκτρέφονται εδώ και δύο γενιές σε εχμαλωσία. Συνήθως ε, στην Ευρώπη ε, το είδος ε, πυθίκου που χρησιμοποιείται είναι πολύ δύσκολο να εκτραφεί. Έγιναν κάποιες έρευνες προσπάθειας εκτροφής σε εχμαλωσία των ζώων αυτών αλλά δεν ήταν επιτυχής οι δοκιμές αυτές. Ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων είναι λιγότερο από το 20% των ε, ζώων που χρησιμοποιούνται ε, στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Κανένας ε, δεν έχει αποδείξει ότι είναι δυνατόν να εκτραφούν αρκετά ζώα δεύτερης γενιάς για, για τα πειράματα μου φαίνεται λοιπόν ε, πολύ άσοφη μία πρόταση που να απαιτεί ε, χρήση συγκεκριμένου είδους ζώου τη στιγμή που δεν ε, υπάρχει απόδειξη ότι υπάρχουν αρκετά τέτοια ζώα. Προτείνω λοιπόν να διαγραφεί η διαταξή αυτή ή τουλάχιστον αποτελεί αντικείμενο μελέτης σκοπιμότητας. Δηλαδή να πρέπει να συμμορφωθούμε τη διάταξη αυτή εάν είναι δυνατόν. Εάν όχι, εάν αφήσουμε τη διάταξη αυτή ως έχει, τότε προφανώς ε, θα αυξήσει πάρα πολύ το κόστος των ζώων αυτών, θα αυξήσει την αβεβαιότητα, διότι θα είναι αδύνατο να βρεθούν τα ζώα για τις έρευνες ε, και το αποτέλεσμα θα ήταν ότι κανένας δεν θα αναθέτει πια τέτοιου τύπου έρευνε εντό τη Ευρώπη. Ε, άρα οι έρευνε αυτέ θα μεταφερθούν σε άλλε χώρε, προφανώ στις Ηνωμένε Πολιτείε, τη Ιαπωνία, την Ινδία και την Κίνα. Κύριε Πρόεδρε, τα ίδια ζώα θα χρησιμοποιηθούν ε, στα ίδια πειράματα σε, άλλα ζώα, σε άλλες χώρες ε, όπου οι ε, ε, ε, διατάξεις για την προστασία των ζώων είναι λιγότερο αυστηρές. Και η Ευρώπη και τα ζώα θα υποφέρουν από αυτό. θα είναι εις βάρος και της Ευρώπης και των ζώων. Και το τρίτο πρόβλημα είναι στη διάταξη 16 που έχει να κάνει με την επανάχρηση των ζώων. Συνήθως τα ζώα χρησιμοποιούνται μία φορά. Ε, συνήθως ένα ζώο ισούται με ένα πείραμα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου οι δοκιμές ε, απαιτούν ε, ιδιαίτερα πολύπλοκη ε, εκπαίδευση ή πολλή προετοιμασία πριν να μπορεί να διεξαχθεί το πείραμα. Να σας δώσω ένα πείραμα που γνωρίζω καλά. Εάν μελετάει κανείς τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος ενός ε, πυθικοειδού, ε, θα πρέπει να τα εκπαιδεύσει. Ε, κάτι τέτοιο θα ήταν να χρησιμοποιούμε μια οθόνη touch screen υπολογιστή και όταν ε, πετύχει τη σωστή σειρά ο τότε τον ανταπίβουμε με φαγητό. Ε, τέτοια εκπαίδευση μπορεί να διαρκέσει έξι μήνες ή περισσότερο. Το ίδιο όμω το πείραμα μπορεί να διαρκέσει τρει μέρε. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ε, πρόκειται για μια ήπια, εκπαίδευση του, ε, ήπια μεταχείριση του ζώου. Έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο ζώο αρκετέ φορέ, γιατί δεν έχει νόημα ε, να εκπαιδεύουμε το ζώο έξι μήνε για άλλη φορά. Αν το κάνουμε αυτό, θα αυξήσουμε τον αριθμό των επιθήκων που θα χρησιμοποιούμε για τα πειράματα αυτά. Άλλο παράδειγμα είναι στα τροκτικά. Εάν θέλουμε να παρακολουθήσουμε την, ε, τα επίπεδα ορμόνης ε, ή την ε, πίεση του αίματός τους, δεν θέλουμε να πάρουμε δείγμα αίματος, διότι αυτό δημιουργεί αγωνία στο ζώο και έτσι και έτσι ε, βγαίνουν λανθασμένα τα αποτελέσματα. Οπότε τι κάνουμε. Εμφυτεύουμε ένα ε, τσιπ ε, όταν το ζώο είναι ανέστητο, το οποίο παρακολουθεί ε, τα επίπεδα ε, πίεσης του αίματος ή ορμόνης. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να καταχωρεί όλα τα... όλα τα στοιχεία που θέλει παρακολουθώντας αυτά που μεταδίδει αυτός ο μικρός πομπός. Ε, όσον αφορά την προστασία των ζώων, λοιπόν, ε, έχει πολύ περισσότερο νόημα να χρησιμοποιούμε ε, το ε, ίδιο ζώο σε, πολλά, σε πολλές δοκιμές. Σύμφωνα με το κείμενο εδώ πέρα, όμως επιτρέπεται να ξαναχρησιμοποιήσουμε τα ζώα σε δοκιμές μόνο σε περίπτωση που η δεύτερη είναι η ιδιαίτερα ήπια μορφή δοκιμής. Καταρχήν θα πρέπει να ορίσουμε το πόσο ήπιο ή μη είναι ένα πείραμα πριν τη δοκιμή ε, και αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα σταματήσει οποιαδήποτε επανάχρηση ζώων στις, ε, ε, στις εμελιώδεις έρευνες. Έτσι, οι έρευνες θα διαρκέσουν περισσότερο, θα στοιχίζουν περισσότερο, ο αριθμός ζώων που θα χρησιμοποιούνται στις δοκιμές θα αυξηθεί σημαντικά συμπεριλαμβανομένου του, αριθμού ε, και γενικά θα αυξηθεί και για πάρα πολύ η γενική ταλαιπωρία των ζώων, η συνολική ταλαιπωρία των ζώων. Μου φαίνεται ότι η σύνταξη της ε, συγκεκριμένη ε, διάταξη δεν πετυχαίνει κανέναν από του στόχου τη. Ε, κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι το δεκάλεπτό μου τελειώνει. Ε, Αυτά τα τρία θέματα που ανέφερα είναι οι προτεραιότητες για τη θεμελιώδη έρευνα για τους ακαδημαϊκούς ερευνητές. Σε περίπτωση που η Επιτροπή σας μπορέσει να αντιμετωπίσει τα τρία αυτά ζητήματα, θα διασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την θεμελιώδη γιατρική έρευνα στα πανεπιστήμια και τα, και τα κέντρα έρευνα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε με ερωτήσεις σε λίγο. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας ε, τώρα. Τον λόγο έχει ο δόκτωρ Φελίπε Ντετίο. Συγγνώμη που δεν μπορώ να προφέρω το όνομά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω τα, την παρουσίασή μου στα γαλλικά. Αλλά βεβαίως μπορώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση στα αγγλικά. Εγώ είμαι κτηνίατρος, είμαι υπεύθυνο της ανεφαβέντης ε, του τμήματος που, αφορούν που ασχολείται με την τοξικολογία, δηλαδή με την ε, ε, με τον αντίκτυπο ενός ε, φαρμάκου. Μιλάω ως εκπρόσωπος Άννεφ Αβέντης, αλλά νομίζω ότι ένα τμήμα τη Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία, συμφωνεί μαζί μου. Είναι μία από, τις μεγαλύτερες, από τους μεγαλύτερους όμιλους ε, ε, φορείς έρευνας φαρμακευτικής, ε, πρώτη μάλιστα στην έρευνα για τον εμβολιασμό. Επίση, είμαστε πολύ παρόντε ε, στι αναδιόμενες, ε, τις αποκαλούμενες αναδιόμενες χώρες, όπου τα, όπου τα ζητήματα της δημόσιας υγείας είναι πολύ σημαντικά και αποτελούν και προτεραιότητα όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση. Μιλάμε για την αναθεώρηση μιας οδηγίας ε, κοινοτικής που είναι ε, μια ε, ένας χρυσός κανόνας στην δουλειά μας. Εμείς σε εργαστηριακό επίπεδο χρησιμοποιούμε τα ζώα όχι ως αυτό σκοπό αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε καινοτόμα φάρμακα αποτελεσματικά και ε, βεβαίως ασφαλή ε, φάρμακα που τοποθετούνται στην αγορά για τους ε, συμπολίτες μας. Τρία τέταρτα των φαρμάκων παράγονται στην Ευρώπη και η αξιολόγησή τους γίνεται στην Ευρώπη. 80% της ε, έρευνας και της ανάπτυξης εμβολίων γίνονται με τη χρήση ανώτερων θηλαστικών και άλλων ζώων και ένα πολύ μεγάλο τμήμα γίνεται και στη Γαλλία. Γνωρίζουμε πολύ καλά και εφαρμόζουμε τον αρχή των τριών R, ε, αναπαραγωγή, μείωση και βελτίωση, αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση. Όταν υπάρχει μία μέθοδο in τη χρησιμοποιούμε και στο screening ε, για να διαλέξουμε το μόριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και στον άνθρωπο, αλλά πριν πρέπει να ε, επιβεβαιώσουμε ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο. Είναι σαν να ψάχνουμε το κλειδί που θα ε, ανοίξει την συγκεκριμένη κλειδαριά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το κλειδί αυτό δεν πρόκειται να ανοίξει και άλλε κλειδαριέ και αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα. Όταν μιλάμε για την τοξικότητα ενός συγκεκριμένου φαρμάκου, έχουμε τη γενετική τοξικότητα, δηλαδή σχέση μορίου με το DNA, 80% αυτό γίνεται in vitro. Και όταν υπάρχει τέτοια μέθοδος, τη χρησιμοποιούμε. Έχουμε μεθόδους ε, για να παρακολουθούμε τα ε, μόρια, για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, ε, να μην δημιουργήσει μέχρι και θάνατο να μην προκαλέσει μέχρι και θάνατο. Είναι κάτι που είδαμε προσφάτως σε μερικές περιπτώσεις. Δηλαδή το συγκεκριμένο μόριο ε, και η εξέταση του συγκεκριμένου ε, ε, μορίου κατά 80% μπορεί να γίνει με προσωμείωση εργαστηριακά για τον άνθρωπο αλλά για το υπόλοιπο 20% πρέπει να περάσουμε από το ζώο. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις βασικές πτυχές ε, της πρόταση αναθεώρησης οδηγίας, ε, για, στις οποίες θα ήθελα να επιμείνω. Πρώτον, ο συνάδελφο Μάτφιλ το ανέφερε ήδη, περιορισμός ε, της ικανότητας των ερευνητών χρήσης των ζώων σε εργαστηριακές συνθήκες στην Ευρώπη και ειδικότερα των ανώτερων θηλαστικών των Ε, τότε μιλώντας βέβαια για τις πιο εκφυλιστικές ασθένειες ε, των, ε, που πλήττουν τους ανθρώπους, ε, η τοξικολογία είναι μία από τις μεθόδους που δημιουργεί οδύνη στα ζώα. Αν δεν γίνουν κάποιες έρευνες, κάποιες δοκιμές σε πυθίκους, δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει η φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη. Πρέπει να περάσουμε από τα ζώα γιατί δημιουργούνται αντισώματα ε, σε φάρμακα ε, για ανθρώπινη χρήση. Ε, δεν δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να ελέγξουμε το μακροχρόνιο αντίκτυπο ενός φαρμάκου. Γιατί μερικά στοιχεία υπάρχουν δυστυχώς μόνο στον πίθηκο. Τώρα, ε, τα το επώδυνο πρωτόκολλο που θα μπορούσε να απαγορευτεί, μιλάμε για το άρθρο 15 Έρευνα δηλαδή για τα νέα εμβόλια που έχουν να κάνουν με τις οικές ασθένειες, τις ιογενείς ασθένειες. Ε, οι έρευνες αυτές και οι δοκιμές μπορούν να γίνουν μόνο στα πυθικοειδή, ε, γιατί μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ανάπτυξη ενός όγκου, για παράδειγμα στο ζώο, ε, μακροπρόθεσμα ομοιάζει με την αντίστοιχη στον άνθρωπο. Άρθρο 37. Σωστή αξιολόγηση της σχέσης κόστους και αποτελεσματικότητας της έρευνας. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου, όταν βρισκόμαστε Είμαστε σε εφαρμοσμένη βέβαια έρευνα πάντοτε ο μακροπρόθεσμος στόχος, το μακροπρόθεσμο όφελος δεν είναι εμφανής από την αρχή. Οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Ας πούμε, αναπαραγωγικές ασθένειες, πρέπει να περάσουμε από τα πυθικοειδή. Είναι κάτι ε, το οποίο και πάλι δυστυχώς ομοιάζει με ε, τον άνθρωπο. Ε, μιλάμε και για ξενιστές αλλά και για δότες. Όλα αυτά αφορούν βεβαίως και τη μεταμόσχευση οργάνων. Κάτι ακόμη, σε αυτά τα άρθρα υπάρχουν ορισμένες ιδέες που εγώ θεωρώ εσφαλμένες. Μπορεί να, υπάρχουν και, μπορεί να δημιουργήσουν ένα αρνητικό αντίκτυπο ε, στην προστασία των ζώων. Ε, αναφέρθηκε ας πούμε ο συνάδελφος προηγουμένως στο εξής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ε, ένα ζώο υπάρχει στη φύση, τότε ο κωδικός μας εμάς είναι F μηδέν εμπροκειμένο. Μπορεί να είναι οπουδήποτε, στην Κίνα, στην Καμπότζη, οπουδήποτε. Το να το πιάσουμε λοιπόν το ζώο από τη, στη φύση ε, σημαίνει ότι μειώνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους. Τότε λοιπόν φτάνουμε στα ζώα F1, τα ζώα τα οποία δεν, έφτασαν, δεν γνώρισαν ποτέ την ελευθερία της ε, άγριας ε, φύσης, ε, και οι περισσότερες ε, φαρμακευτικές εταιρείες τέτοια ζώα χρησιμοποιούν. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ε, το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι καμία χώρα, κανένα εργαστήριο δεν ήταν σε θέση, μιλάω ας πούμε η δική μου περίπτωση, ε, για τον πίθηκο, κανένας δεν μπόρεσε να φτάσει στα ζώα F2. Για να γνωρίζουμε λοιπόν Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ότι ο πίθηκος ε, έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό θηλυκών από ό,τι αρσενικά και επομένως ας πούμε ένα αρσενικό 25 θηλυκά όμως ένα ε, φάρμακο πρέπει να δοκιμαστεί και σε αρσενικά και σε θηλυκά οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να δημιουργεί ένα πρόβλημα επανάχρηση που ανέφερε και ο συνάδελφος, το άρθρο 16. Θέλουμε να είναι η ελάχιστη δυνατή, όπως εξηγίζει ο Μάρκ, εμείς χρησιμοποιούμε ζώα στα οποία έχουμε εμφυτεύσει μία συσκευή που μας επιτρέπει εξ αποστάσεως να ελέγξουμε ε, την ε, πίεση ε, του αίματος, το κάνουμε αυτό ακόμη και στο σκύλο και μπορούμε να το κάνουμε και στον πίθηκο. Αυτή η διαδικασία, ε, η χειρουργική δηλαδή εμφύτευση ενός, ε, μιας τέτοιας συσκευής σε ορισμένες ε, χώρες θεωρείται ότι είναι επώδυνη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κάτι ακόμη το οποίο θα αναφέρω και αργότερα, θα ήθελα ήδη να πω ορισμένα πράγματα, είναι το γραφειοκρατικό άχθος μπορεί να δημιουργήσει βέβαια και πιο συγκεκριμένους κινδύνους. Μια επιτροπή διοντολογίας είναι κάτι το οποίο και εμείς επιζητούμε. Μια αρμόδια αρχή δηλαδή σε κάθε κράτος μέλος, γιατί πιστεύουμε ότι ο καλύτερος έλεγχος που μπορούμε να έχουμε επί της έρευνας είναι αυτός που γίνεται επί τόπου από τους ε, εμπλεκόμενους επιστήμονες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και επιπλέον έλεγχοι η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και περίπου 20 χρόνια. Πρόκειται για επιτροπές ε, κάθε ερευνητικού ιδρύματος, στο, στην οποία συμμετέχουν ερευνητές, ε, αλλά και έχουν και ε, μέλη τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ερευνητική διαδικασία. και αυτό νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, οι αιτήσιε επιθεωρήσεις είναι κάτι το οποίο επίσης δημιουργεί πρόβλημα. Ούτως ή άλλως υπάρχει πολύς έλεγχος ε, ε, για την καλή εργαστηριακή πρακτική. Υπάρχει έλεγχος κάθε δύο χρόνια. Ούτως ή άλλως ε, υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης του εργαστηρίου από πιστοποιημένους ε, ελεγκτές εξουσιοδοτημένους ελεγκτές. Ε, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ένας επιπλέον έλεγχος σε, αυτήν την ετήσια, σε αυτόν τον ετήσιο έλεγχο. Ούτως ή άλλως τακτικός έλεγχος ε, πολύ διεξοδικός γίνεται κάθε δύο χρόνια και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ελέγχουμε πλήρως ε, την κατάσταση στην φαρμακοβιομηχανία. Κάτι ακόμη να, και να ολοκληρώσω γιατί... Τελειώνει και ο χρόνος μου. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την έρευνα στην Ευρώπη και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί ε, με τις διατάξεις που μπορεί να επιτρέψουν μετάβαση σε άλλες χώρες της Ασίας για παράδειγμα. Εκεί τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά, δεν συμφωνούν πάντοτε με τις οδηγίες ε, τις οποίες ε, εμείς υποστηρίζουμε εδώ στην Ευρώπη όσον αφορά την ασφάλεια των φαρμάκων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην τρίτη εμπειρογνώμονα, την κυρία Πένι Χόκκινς, αναπληρώτρια διευθύντρια του, του, ε, του τμήματος ζώων που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. Εγώ εκπροσωπώ το Eurogroup. Καλωσορίζουμε την ε, οδηγία αυτή θεωρούμε ότι ε, επιτυχάνεται σημαντική πρόοδος για όλα αυτά τα θέματα από την αρχική σύνταξη της οδηγίας και έχει αλλάξει και η κοινή γνώμη, η άποψή της για τα θέματα αυτά. Επομένως η νομοθεσία πρέπει να λάβει υπόψη της την καινούργια αντίληψη της κοινή γνώμης αλλά και της καινούργιες ε, απόψει των επιστημόνων από το 1986 και μετά. Οι επιστήμονες δεν εργάζονται ε, σε ένα ηθικό κενό, είναι υπόλογοι στην υπόλοιπη κοινωνία. Το Eurogroup πιστεύει ότι η καινούργια πρόταση οδηγίας έχει πολύ σωστές αρχές, αλλά έχουμε και κάποιες ανησυχίες, τις οποίες θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω συνοπτικά. Ε, να πω καταρχάς ποιες είναι οι θετικές εξελίξεις. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής και περιλαμβάνει περισσότερους επιστημονικούς σκοπούς, περισσότερα επιστημονικά είδη και ούτε καθεξής. Βασική έρευνα, πανεπιστημιακή έρευνα σε κεφαλόποδα, σε εμβριονικά ζώα, σε ζωικά έμβρια και το καθεξής. Θα πρέπει να ρυθμίζονται σωστά όλα τα θέματα που προκαλούν οδύνη. Το θέμα της οδύνης θα πρέπει να καλύπτεται ανεξαρτήτως είδους ή στάδιο της εξέλιξης. Στηρίζουμε την σαφέστατη απέτηση προς τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή όλων των περιορισμών. Όλοι, όλα αυτά είναι θεμελιώδη για οποιοδήποτε τέτοιου είδους νομοθεσμισία. Η αντιακατάσταση των ζώων πρέπει να είναι προτεραιότητα και θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για τα τρία ρο, το replacement δηλαδή την αντικατάσταση και για τις καλές πρακτικές και για την επικύρωση ε, μέσω των ε, προτύπων επιβεβαίωσης όλων αυτό. Θα πρέπει η διαδικασία έγκρισης να είναι πολύ ε, ισχυρή, σταθερή σε οποιοδήποτε χρησιμοποιεί η έρευνα πάνω στα ζώα. Έχουμε ένα σύστημα έγκρισης και εξουσιοδότησης τριών επιπέδων, το οποίο λειτουργεί πολύ σωστά στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 86 χωρίς να υπάρχουν ε, προβλήματα στην επιστημονική δραστηριότητα. Σημαντικό είναι το θέμα της κατάρτισης και της απόδειξης των επιστημονικών προσόντων. Πολύ θετικό είναι το ότι πρέπει να εξετάζεται και η ηθική σκοπιά κάθε προγράμματος. Η ηθική αξιολόγηση δηλαδή από την αρμόδια αρχή, από τα τοπικά σώματα ηθικής και δεντολογίας, αλλά και από τις Εθνικές Επιτροπές για την Καλή Διαβίωση των Ζώων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν στην οδηγία και δείχνει η οδηγία ότι λαμβάνει υπόψη της όλα τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα για να μειωθεί η οδύνη των ζώων. Έλλειψη πληροφόρησης. Μεγάλη ανησυχία αυτή για το Eurogroup. Καλωσορίζουμε λοιπόν την ε, απέτηση αυτή να δημοσιεύονται ετήσια στατιστικά στοιχεία για όλα αυτά τα θέματα και καλωσορίζουμε και τη δημοσίευση περιλήψεων, μη τεχνικών περιλήψεων για τα θέματα αυτά, για τις επιστημονικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται. Το καινούριο παράρτημα 4 βασίζεται στο παράρτημα 8 της Σύμβασης ETS 123 του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό και έχει γίνει μετά από πλήρη διαβούλευση με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ωστόσο, παραμένουν κάποιες ανησυχίες από πλευράς μας για όλα αυτά τα θέματα. Θα επανέλθω αργότερα. Εμείς ε, είμαστε υπέρ των περιορισμών των μη ανθρωπίνων πρωτογενών θηλαστικών και είναι σημαντικό να μειωθεί η οδύνη των πρωτογενών θηλαστικών. Το Eurogroup θεωρεί λοιπόν ότι πολλές από τις αρχές της πρότασης είναι θετικές. Ωστόσο κάποια άρθρα είναι αμφίσιμα, δυσνόητα. Το άρθρο 2 στο πεδίο εφαρμογής λέει ότι η οδηγία δεν θα ισχύσει σε επεμβατικές ερευνητικές μεθόδους. Επεμβατικές με τη χειρουργική έννοια του όρου. Υπάρχουν διάφορες άλλες ε, ε, έννοιες που μπορούν να προκαλέσουν οδύνη στα ζώα. Κάποια άλλα άρθρα είναι πολύ περιορισμένα, θα πρέπει να πάνε πολύ πιο πέρα. Μας ανησυχεί το θέμα της ευθανασίας των αναλλακτικών ε, μεθόδων ως προς τα πρωτογενή θηλαστικά και ούτω καθεξής. Και στο παράρτημα minimum standard και όχι best practices και όχι καλές πρακτικές. Αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερο, το κείμενο πρέπει να ξαναμπεί στο παράρτημα γιατί περιλαμβάνει πολύ σημαντικά στοιχεία για την βιολογία και τη συμπεριφορά των ζώων και έχουμε λεπτομερείς κατευθυντήρες γραμμές εκεί. Και τρίτο, πολύ, μεγάλος, ε, πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο δίδεται. Δηλαδή το 2012 θα αναθεωρηθούν τα, η νομοθεσία για τα, τα λαγόμορφα και το 2017 για τα κοινοειδή. Ε, πάρα πολλά χρόνια δηλαδή αυτά θα περάσουν πριν υπάρξει ενδιάμεση αξιολόγηση. Έχουν περάσει άλλα δύο χρόνια από την τελευταία φορά που είχαν προσκληθεί να πούν την άποψή τους και οι εκτροφείς και διάφοροι εκπρόσωποι των διαφορομένων ομάδων. Δεν πρέπει να σημειωθούν άλλες καθυστερήσεις. Τώρα, ως προς την σοβαρότητα, το σύστημα ταξινόμησης των, της σοβαρότητας πρέπει να υπάρξει και να γίνεται ιεράρχηση. Δεν είναι σαφή όλα αυτά. Πρέπει οι ορισμοί να γίνουν πολύ πιο σαφείς του τι σημαίνει μέτριο ή μετριασμένη επέμβαση ή μη μετριασμένη διότι πολλά άρθρα εξαρτώνται από την ταξινόμηση και τους ε, εκάστοτε ορισμούς. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής περίληψης για ήπια project όταν δεν χρησιμοποιούν μη ανθρώπινα πρωτογενή θηλαστικά. Αυτό είναι λάθος. Ο κάθε οδύνη ζώου είναι σημαντική και οι φορείς ενδιαφέρονται για την οδύνη όλων των ζώων. οι περιορισμοί στους σκοπούς που επιτρέπονται είναι σημαντικοί αλλά όχι αρκετοί. Η επιστημονική κοινότητα, η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει πει επανειλημμένως ότι δεν τις χρησιμεύουν τα μη πρωτογενή θελαστικά στην έρευνα. Ευκαιρία λοιπόν να τα σταματήσει να τα χρησιμοποιεί και να το δείξει αυτό. και τα 7 ή 10 χρόνια του παραρτήματος 3 ε, για τα ζώα F2 είναι ένα χρονικό διάστημα που θα πρέπει να αλλάξει και να διαγραφεί η ρήτρα προφύλαξης. Άλλωστε έχουμε και πολύ μεγάλες ανησυχίες για τη χρήση των μεγάλων ε, πυθίκων, Great Apes. Τώρα για τα θέματα της ευθανασίας. Να δεν συμπεριλαμβάνονται και τα σπόνδυλα. Έχουμε νευρομυϊκούς παράγοντες δέσμευσης. Έχουμε θανάτωση τροκτικών με άλγων. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν οδύνη στα ζώα. Πρέπει να βελτιωθεί η διατύπωση του κειμένου. Το Eurogroup επίσης ε, θεωρεί ότι είναι σημαντικό ότι προβλέπονται εναλλακτικέ μέθοδοι στην πρόταση οδηγίας. Τα εθνικά εργαστήρια πρέπει να βοηθήσουν την ΕΚΒΑΝ. Όχι όμως ε, μόνο στις τοξικολογικές δραστηριότητες, γιατί είναι λίγες αυτές οι τοξικολογικές διαδικασίες. Χρησιμοποιούνται ζώα και για άλλους σκοπούς και με άλλες εναλλακτικές μεθόδους. Θα πρέπει η οδηγία λοιπόν ρητός να αναγνωρίσει την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών μεθόδων σε όλους τους επιστημονικούς τομείς ε, ερευνητικής ή δραστηριότητας πανεπιστημιακής ημί. Θεωρούμε ότι πολλές από τις αρχές ε, υπάρχουν στην οδηγία, αρχές που θα πρέπει να διέπουν τα πειράματα σε ζώα, ωστόσο κάποια σημεία του κειμένου αποτελούν πλήγμα διότι συμβάλλουν στη μεγάλη οδύνη των ζώων. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των οργανώσεων για την προστασία των ζώων και έχουμε τα τρία ρότα περιβόητα και την αποδοχή του ότι είναι πολύ σημαντική η καλή ε, προστασία και η καλή διαβίωση των ζώων. Τα τρία ρότα στα αγγλικά τα οποία σημαίνουν αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση. Είχε, έχει έρθει η ώρα να βελτιωθεί η νομοθεσία η οποία ήταν πολύ απαξιωμένη, πολύ παλιά και θα, το καινούργιο κείμενο είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερες συνθήκες στον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Με έχουν προσεγγίσει και ο οργανώσεις ασθενών. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σόφια Πιτετζήμεν που, είναι, που εκπροσωπείται την ε, Ένωση ε, ε, Ιατρικών Φιλανθρωπικών Ενώσεων. Σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο να συμμετάσχω στη συζήτηση σήμερα. Η Ένωσή μας είναι οργάνωση που εδρεύει στις, στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετέχουν σε αυτήν περίπου 150 φιλανθρωπικά ιδρύματα που χρηματοδοτούν τις ιατρικές έρευνες. Από πολύ μεγάλες ε, οργανώσεις συμμετέχουν ε, μέχρι πολύ μικρές, ε, στις οποίες συμμετέχουν κυρίως ασθενείς. Ένα ε, όμως είναι το κοινό θέμα. Τους ενδιαφέρει η ε, ευημερία των ασθενών. Μόνο το 1 τρίτο των οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ένωσή μας ε, χρηματοδοτούν ανα πάσα στιγμή ε, πειράματα σε ζώα. Στηρίζουν όμως το θέμα αυτό διότι είναι σημαντικό για τους, ασθενεί, για τους ασθενείς. Ε, σχεδόν όλες οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού του, του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να δεχτεί τα πειράματα στο ζώα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις και εφόσον ε, ε, διαξάγονται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ε, και άλλωστε όλα αυτά θεσπίζονται στο νόμο. Ε, εξετάσαμε το σχέδιο της οδηγίας. Ε, δεν ε, θα μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά την αύξηση της γραφειοκρατίας ή, ή τον περιορισμό των δοκιμών ε, που θα είναι τελικά εις βάρος ε, των ασθενών. Άλλωστε θα μπορούσαμε να έχουμε αύξηση της γραφειοκρατίας ε, χωρίς πειράματα σε ζώα. Αυτό θα ήταν η χειρότερη δυνατή περίπτωση. Θα ήθελα σήμερα να σας δώσω παραδείγματα των οφελών για τους ασθενείς από τα πειράματα σε ζώα και γιατί τα υπερασπιζόμαστε. Για παράδειγμα, έρευνες για το εγκεφαλικό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ε, τροχτικά και γάτες. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται. Ανεσυτοποιείται το ζώο και ουσιαστικά μιμούμαστε τη διαδικασία που ε, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ε, ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Δηλαδή ουσιαστικά μπλοκάρουμε μια αρτηρία. Αυτό γίνεται στο εγκεφαλικό χωρίς ε, να, ε, ξανα, ε, χωρίς να ανακτήσει την συνείδησή του το ζώο μπορούμε να το σκοτώσουμε, να του κάνουμε ευθανασία και να εξετάσουμε το τι γίνεται στον εγκέφαλό του. Σε κάποια από τα πειράματα μπορούμε επίσης Ε, να χορηγήσουμε στο ζώο κάποιο ε, νευροπροστατευτικό ε, μέσο το οποίο προστατεύει το ζώο και έτσι βλέπουμε τι γίνεται στο ζώο στο μικροσκόπιο. Βλέπουμε δηλαδή ζωντανά κύτταρα και όχι τα νεκρά κύτταρα που που ε, ε, οδηγούν στα συμπτώματα της, του εγκεφαλικού επεισοδίου στους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ζώα. Για να καταλάβουμε το τι πάει στραβά σε έναν άνθρωπο και το τι ε, ουσίες πρέπει να του χορηγηθούν, ε, πρέπει να έχουμε τις ίδιες αρτηρίες, εγκεφαλικά κύτταρα, καρδιά κτλ. Ο πατέρας μου ε, αυτή τη στιγμή ε, περνάει ε, από στατική θεραπεία μετά από δύο σημαντικά εγκεφαλικά. Είναι πια πολύ αργά. για αυτόν ε, μόλις ε, έγινε 80 ετών, ε, του άρεσε να περπατάει πολύ, παίζε σκουός και έκανε σκι. Τώρα πια δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Τελευταία φορά που ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουν μαζί με έναν κύριο που τον λένε Μάικλ Ρόμπινς, ο οποίος έχει Πάρκινσονς. Είμαι βέβαια ότι γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει. Οι νευρώνες στον εγκέφαλο δεν επικοινωνούν πια μεταξύ τους, κάτι που έχει επιπτώσεις στην κινητήρια ικανότητα του ανθρώπου αλλά και σε πολλές άλλες λειτουργίες. Ήταν τόσο ε, κακή κατάστασή του που η, γυναίκα, η γυναίκα του και τα παιδιά του ε, δεν ε, μπορούσαν να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο μαζί του όταν διάβαζε εφημερίδα διότι ε, έτρεμε τόσο πολύ που έκανε πάρα πολύ θόρυβο. Του πρόσφεραν μια θεραπεία που λέγεται Deep Brain Stimulation. αυτό εμφυτεύει ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο και έτσι ανακουφίζει τα συμπτώματα όταν ε, ανάβει κανείς ε, τη συσκευή, ο Μάικλ Ρόμπινς λειτουργεί ακριβώς όπως ε, εγώ και εσείς. Μόλις κλείσει η, η συσκευή αυτή, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Περίπου 20 επίθηκοι έχουν χρησιμοποιηθεί για τα σχετικά πειράματα και 40.000 άνθρωποι έχουν υποφεληθεί από τη, ε, από τη θεραπεία αυτή. Ε, πολύ δικαιολογημένα οι δοκιμές σε πρωτεύοντα θηλαστικά δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες, ε, αλλά ε, τα ωφέλη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δύο φωτογραφίες, δύο περιστατικά σας ανέφερα, αλλά σκεφτείτε οποιαδήποτε ε, γιατρική ε, θεραπεία, ε, μεταμόσχευση καρδιάς ή αλλαγή του κερατοειδούς. Θα την κάνατε ή θα αφήνατε τα παιδιά σας να το κάνουν, αν δεν είχε δοκιμαστεί πριν, αν δεν αν δεν είχαν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα βρετανικά πρότυπα που απαιτούν ότι πρέπει να δοκιμαστούν ε, οι θεραπείες αυτές σε ε, τουλάχιστον ε, δύο θηλαστικά εκ των οποίων το ένα δεν θα πρέπει να είναι τροφικό. Θα γνωρίζαμε πώ αντιδράει το σώμα στην ασθένεια, τι ακριβώ πάει στραβά κτλ. εάν δεν κάναμε δοκιμέ σε ζώα. Πρόσφατα μίλησα με έναν ερευνητή ο οποίο χρησιμοποιεί νηφίτσες. Ε, είναι ε, τα μόνα ζώα που έχουν ε, το, το, ίδιο αντανακλαστικό εμετού με τα με τους ανθρώπους. Γιατί χρησιμοποιεί τέτοια ζώα για να εξερευνήσει τα, ε, ε, ε τις αντιδράσεις ε, του, ε, οργανισμού, του ανθρώπινου οργανισμού στη χημειοθεραπεία για τον καρκίνο. μίλησα πρόσφατα με μια γυναίκα και την κόρη της. Η κόρη της ήταν ε, έγκυος. ο γιατρός μου είπε ότι χωρίς τα αντιεμετικά που είχαν δημιουργηθεί πάνω στις νηφίτσες που επέτρεπαν τη συνέχιση της χημειοθεραπείας Σκοπίας Ούτε αυτή, ούτε η κόρη της θα μπορούσε να συνεχίσει τη θεραπεία καρκίνου που ε, περνούσαν. Ε, νομίζω ότι έχουμε λοιπόν ε, πολύ σαφή ωφέλη από την έρευνα αυτή. Η μητέρα μου πέθανε από καρκίνο πριν 10-11 χρόνια και όταν πέθανε γνώριζα ότι θα ήμουν διατεθειμένη να υπερασπιστώ το δικαίωμα των ερευνητών να αναπτύξουν τα φάρμακα που θα μπορούσαν να την ανακουφίσουν, όπως άλλωστε κάνω σήμερα. Κανένας δεν θέλει να χρησιμοποιήσει ζώα σε ε, επιστημονικές έρευνες. Ε, δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς ε, άδεια να το κάνει εάν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις ή λιγότερο βάναυση τρόποι. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στα, σε εναλλακτικέ λύσεις διότι αναφέρεται συχνά αυτό. Περίπου τρία, πριν τρία χρόνια μια οργάνωση ήρθε και μου μίλησε για εναλλακτικέ λύσεις, μοντέλα υπολογιστών κλπ. Ε, πολύ χρήσιμα μέσα αυτά. Και τους είπα ότι αν μου πείτε πώς μπορείτε να μιμηθείτε ένα ε, ζωντανό ανθρώπινο σώμα όπως τα παραδείγματα που σας ανέφερα νωρίτερα για να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες θα συμμετάσχω στην εκστρατεία σας και το εννοούσα. Μου απάντησε ναι είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Τρία χρόνια έχουν περάσει ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση από την οργάνωσή του για το πώς ε, μπορούν ε, να κάνουν τη δουλειά που κάνουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις μας. Όταν ο κόσμο δεν είναι ικανοποιημένο με τη δουλειά που ε, χρηματοδοτείται, ε, ε, όπου χρησιμοποιούνται ζώα, το, συνήθως το επιχείρημα είναι ότι είναι ανήθικο. Αυτό όμως ξεχνάει την πραγματικότητα της ασθένειας. Είναι ηθικό το να μην το κάνουμε. Αν μπορούμε να ανακοφίσουμε ε, τον πόνο ανθρώπων ε, χρησιμοποιώντας ε, ζώα για να αναπτύξουμε θεραπείες. Εάν μπορούμε να βρούμε τρόπο πιο γρήγορο, πιο φτηνό, διότι είναι πολύ ακριβά τα πειράματα αυτά, ή πιο αποτελεσματικό, ή εξίσου αποτελεσματικό, τότε θα είμαστε υπέρ. ακούσαμε από τον κύριο Χόκκινς για τα τρία ρο, αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση. Και υπάρχει ανησυχία σχετικά με την αύξηση των αριθμών ε, στις στατιστικές του Ηνωμένου Βασιλείου για τη χρήση των ζώων. Αυτό φαίνεται ότι ε, είναι αντίθετο με την προσπάθεια μείωσης. Ε, το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ζώα εκτρέφονται με γενετικές τροποποιήσεις που θα τα κάνουν καλύτερα πρότυπα για συγκεκριμένες ασθένειες. Η εκτροφή αυτή τη στιγμή στιγμή ε, συμπεριλαμβάνεται στα ποσά, στα, στους αριθμούς αυτούς ε, και γι' αυτό βλέπουμε αύξηση. τα ζώα, αυτά τα εκτροφόμενα αυτά ζώα θα είναι καλύτερα πρότυπα για τις ασθένειες. Στο μεταξύ θα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, τα υψηλότερα επίπεδα ευζωίας για να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να συνεχιστεί η έρευνα προς όφελος των ασθενών. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι με ενδιαφέρει ε, το συμφέρον των ασθενών, αλλά ε, το 90% των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ε, στα ζώα αναπτύχθηκαν ουσιαστικά για ανθρώπους. Έτσι λοιπόν φωλούνται και τα ζώα από τις έρευνες αυτές. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι οι ομιλητές ε, συμφωνούν ότι είναι ένα ηθικό δίλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι υπάρχει στην οδηγία, να δούμε τα διάφορα άρθρα. Εγώ θα επανέλθω με ορισμένες ερωτήσεις, αλλά καταρχάς ο Γκρέφε Τζουμπάριντορφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν συναντηθήκαμε με τις θρησκευτικέ ομάδες που απαιτούσαν ελευθερία για την άσκηση της ασκίας τους. Τώρα ακούσαμε και πάλι μια πολύ θρησκευτική ομιλία. Μια ομιλία με πάθος. Διότι αν δεν είμαι υπέρ των ασθενών, είμαι αφελής, είμαι ανήθικος και δεν με ενδιαφέρει η ζωή. Μου φαίνεται ότι βρίσκομαι υποπίεση και θα ήθελα να αμυνθώ. Οποιοςδήποτε διαφωνεί δηλαδή, ε, θεωρείται ότι δεν έχει σκεφτεί καλά το θέμα. Όχι, το αρνούμε αυτό. Όσον αφορά την ελευθερία της έρευνας, όπως ακριβώς με την ε, ελευθερία της θρησκείας, θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τεθούν όρια. Ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, ζωντανούς οργανισμούς για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι. Μας ε, λέτε ότι είναι υπερβολικά ρυθμισμένα όλα αυτά και βλέπουμε τώρα ακόμα περισσότερη ρύθμιση. Βρήκα αρκετά μετριοπαθή όμως ε, την ομιλία της ε, εκπροσώπου για ε, την προστασία των ζώων. Δεν μας είπαν ότι θα πρέπει να γίνονται πειράματα, μας είπε ότι θα πρέπει να θέσουμε όρια. Ή τουλάχιστον θα πρέπει να εξετάσουμε την αναγκαιότητα της ηθικολογίας. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την ε, αναγκαιότητα και τις, ε, και τις ηθικές πτυχές για την προστασία των ζώων. Η τελευταία εκπρόσωπος μίλησε υπέρ των ασθενών, δηλαδή εκ μέρους και της βιομηχανίας. Δεν έχω τίποτα κατά των συμφερόντων της βιομηχανίας, αλλά μας λέτε ότι αν ε, δεν ε, είμαστε υπέρ, τότε θα φύγουν οι βιομηχανίες, θα πάνε στην Αμερική. Άλλος συνάδελφος είπε ε, ότι θα πάνε στην Ασία. Πολλές από τις εταιρείες ούτως ή άλλως πάνε στην Ασία, διότι εκεί μπορούν να παράγουν πιο φθηνά τα προϊόντα τους. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη ρύθμιση ή με τα πρότυπα. Άλλοι νόμοι ισχύουν εδώ. Σε αντίθεση με αυτά που είπαμε πριν, όπου μιλούσαμε για τη σφαγή, πολύ βάρβαρα πράγματα. Εδώ πέρα μιλάμε για περιπτώσεις όπου συνειδητά υποβάλλουμε ζώα σε πόνο. Θα πρέπει να υποφέρουν για να μπορούμε να κάνουμε εμείς πειράματα. Δεν θέλω να βγάλω το συμπέρασμα ότι αυτό δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Θα έπρεπε όμως να αντιμετωπίσουμε ε, το γεγονός αυτό. Και με θυμώνει όταν κάποιοι μου, μου λένε ότι είμαι αφελής επειδή ε, έχει πεθάνει η μητέρα του από καρκίνο. Η ε, ζωή είναι επικίνδυνη. Αργά ή γρήγορα όλοι μας, όλοι μας θα πεθάνουμε. Δεν είμαι κοινικός. Αλλά από αυτό να βγάλω το συμπέρασμα ότι επιτρέπεται να κάνω οτιδήποτε σε κάποιον άλλο ζωντανό οργανισμό μου φαίνεται υπερβολικό. Αν μου πείτε να συμβιβαστούμε, τότε μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό που είπε η, ε, αυτή που είναι υπέρ της προστασίας ε, των ζώων, ε, που δεν είπε ότι πρέπει να διαλέξουμε ή το ένα ή το άλλο, μας ε, είπε να εξετάσουμε τις εναλλακτικέ λύσεις ε, για τα πρωτεύοντα ε, θηλαστικά. Πριν 10-15 χρόνια, Οι εναλλακτικέ λύσει που χρησιμοποιούνται σήμερα ε, δεν ε, ε, θεωρούνταν καν δυνατότητα. Θα ήθελα λοιπόν στους εκπροσώπους της βιομηχανίας να πω ότι όσοι είναι υπέρ της προστασίας των ζώων δεν απέκλεισαν τίποτα, μας είπαν να στο συζητήσουμε το θέμα. Ε, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να κατηγορούμε ένα τον άλλο για λάθος θέσεις. Ε, άλλωστε και εσεί ενδιαφέρεστε για, για το συμφέρον της βιομηχανίας. Ε, θυμώνω λίγο με, με το ύφος αυτό. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε όλοι ευγνώμονες για τις παρεμβάσεις ε, των διαφόρων εκπροσώπων. Εμένα η τελευταία ομιλία της εκπροσώπου των ε, φιλανθρωπικών οργανώσεων μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γιατί πραγματικά μας έδειξε την πραγματικότητα του τι σημαίνει στην πράξη. Του να είμαστε μερικές φορές ορθοί σε όλα αλλά μπορεί έτσι να οδηγούμαστε σε μία θέση την οποία δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Δηλαδή βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Να μην είμαστε απόλυτοι δηλαδή. Βλέπουμε πόσο απόλυτοι είναι αυτοί που είναι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των ζών. Όλο και περισσότερο δεχόμαστε το λόμπινγκ ε, των ε, υπερμάχων της προστασίας ζών σε σχέση με το θέμα αυτό. Κανένας δεν θέλει. Κανένας δεν θέλει εσκεμένο, εσκεμένη οδύνη ε, για τα ζώα. Αντιθέτως, αλλά πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα. Ότι υπάρχει μια ιεράρχηση ανησυχιών τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Κατά τη γνώμη μου το να διευκολύνουμε την ιατρική έρευνα με σκοπό να τελειοποιήσουμε θεραπείες ε, χρονίων ε, ασθενειών έχει την πρώτη θέση σε αυτή την ιεράρχηση. Για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία και βέβαια είναι πολύ σημαντικότερη από την απόλυτη προστασία κατά ε, των πειραμάτων ε, σε ζώα και στα ε, ανώτερα θηλαστικά. Όταν δεν υπάρχει βέβαια άλλη εναλλακτική λύση. Δέχομαι ότι η ιατρική έρευνα που πρέπει να χρησιμοποιήσει ζώα ώστε να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο, να βελτιώσει θεραπείες όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, πρέπει να χρησιμοποιεί ζώα και κατά την άποψή μου δεν είναι μόνο αποδεκτή, αλλά είναι απαραίτητη. Και νομίζω ότι στην αναθεώρηση της ε, οδηγίας πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Ναι, είναι σωστό να ε, βελτιώνουμε τις διατάξεις ε, της προστασίας των ζώων, ε, αντικατάσταση, μείωση, βελτίωση, ναι όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να δημιουργούμε εμπόδια στη βελτίωση της γνώσης, με γενικές απαγορεύσεις, χρήσης ανωτέρων θηλαστικών με υπερβολική ρύθμιση της έρευνας Δεν πρέπει λοιπόν να αποδυναμώνουμε, να αποδυναμώνουμε την απαραίτητη έρευνα, τη θεμητή έρευνα. Μερικές φορές ακούω μερικούς ε, ανθρώπους και αναρωτιέμαι και το έχουμε δει πολλές φορές και σε άλλα θέματα που έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή μας. Λέμε η Ευρώπη ότι πρέπει να είναι ορθή, ε, σε όλα ορθή και να μην ε, επιτρέπουμε πράγματα που συμβαίνουν αλλού ε, στον κόσμο. Αλλά ναι βέβαια, τότε θα κάνουμε την εισαγωγή όλων αυτών των φαρμάκων που είναι το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Πρέπει πραγματικά να έχουμε μία ε, αίσθηση των αναλογιών εν προκειμένου. Αν είναι καλό για την ανθρωπότητα να αποδεχθούμε θεραπείες σε συγκεκριμένες ασθένειες πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να πληρώσουμε ένα τίμημα ένα τίμημα όσον αφορά την ανοχή αυτής της απαραίτητης τουλάχιστον ε, δοκιμής σε ζώα, των πειραμάτων σε ζώα. Κύριε Πρόεδρε, εσείς είστε ο εισηγητής και υποθέτω ότι και εσείς ε, θα προσπαθήσετε να εισαγάγετε αυτήν την ε, ισορροπία στην έκθεσή σας, ότι πρέπει να γίνει μια επιλογή και όταν γίνεται αυτή η επιλογή κανείς δεν θέλει να είναι ούτε απάνθρωπος, ούτε εκδικητικός ε, σε σχέση με τα ζώα. Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά πρέπει να αποδεχθούμε ότι κάποιες επιλογές πρέπει να γίνουν και όταν πρέπει να γίνουν επιλογές, τότε η προστασία της ανθρωπότητας από καλπάζουσες ασθένειες, ε, από εκφυλιστικές ασθένειες, ε, είναι τόσο σημαντική ότι ώστε την επιλογή αυτή που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε ένα βαθμό πειραμάτων σε ζώα. Διαφορετικά, όπως ακούσαμε σήμερα, δεν θα ήμασταν σε αυτήν τη θέση, όπου έχουμε νικήσει ορισμένες ασθένειε, ε, ώστε να έχει μετριαστεί ε, ο αντίκτυπο αυτών των ασθενειών στην ανθρωπότητα. Πρέπει πραγματικά λοιπόν να αναγνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα, ε, όσο και αν είναι δύσκολο να το κάνουμε από ορισμένε απόψεις. Ναι, λέει ο πρόεδρο, αυτό ακριβώ προσπαθώ να κάνω Η κυρία Λεφρονσουάζ είναι η σκιώδη συγγήτρια. Την καλώ να πάρει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Είμαι σκιώδηση συγγήτρια για το θέμα αυτό και με την ιδιότητα αυτή θα ήθελα να σας εκφράσω τις απόψεις μου. Καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τους εμπειρογνώμονες για τις πολύ ποιοτικέ τους παρεμβάσεις. Η συνεισοφορά τους μας φωτίζει ε, για και καταλαβαίνουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε το σχέδιο οδηγίας. Έχω συναντηθεί με διάφορους φορείς που εκπροσωπούν διαφορετικές ευαισθησίες για το φάκελο αυτό. Και πιστεύω ότι το σημαντικό είναι το Κοινοβούλιο να εθετήσει μια ισορροπημένη και υπεύθυνη θέση για το θέμα των πειραμάτων σε ζώα. Εγώ είμαι υπέρ ενός κειμένου το οποίο θα επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει η καλή διαβίωση των ζώων, ενός κειμένου το οποίο θα εγγυάται στην έρευνα τη δυνατότητα να σημειώνει πρόοδο και τώρα και στο μέλλον. Όσο πολιτικοί ηθήνοντες πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ερευνητικής δραστηριότητας βρίσκεται στα βέλτιστα δυνατά επίπεδα, έτσι ώστε οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας να μην παραμείνουν κενό γράμμα και να μην υπάρξει επιβράδυση της προόδου μας. Δεν έχουμε τα μέσα σήμερα, κάτι για το οποίο λυπούμεθα όλοι, να ε, μην επιλέξουμε τα πειράματα σε ζώα. Μακάρι να τα είχαμε και να μην είχαμε ανάγκη τα πειράματα σε ζώα. Ωστόσο, οι επιστημονικές εξελίξεις ε, τα τελευταία χρόνια καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση των νομοθετικών διατάξεων στο θέμα αυτό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η αρχή των τριών Ρο, αντικατάσταση, μείωση, βελτίωση είναι και ένας από τους πυλώνες του κειμένου, ώστε να φαίνεται η σκοπιμότητα χρήσης του κάθε ζώου για επιστημονικούς ερευνητικούς σκοπούς. Δηλαδή, ο σκοπός ο οποίος είναι η έρευνα για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. Όσο οι μέθοδοι μας δεν είναι πολύ αποτελεσματικές, ε, οι υπόλοιποι μέθοδοι μας τόσο δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πάυση ε, τέτοιου είδους ε, πειραμάτων. Θα πρέπει να εξαφανιστούν τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα μεταξύ των κρατών μελών. Είναι επενετέως αυτός ο στόχος. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ε, βρισκόμαστε στην αρένα του παγκοσμίου ανταγωνισμού και θα πρέπει η ευρωπαϊκή έρευνα να είναι σε θέση να προοδεύσει και να σταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η καλύτερη λύση η υιοθέτηση ενός καινούργιου κειμένου περισσότερου δυσμευτικού το οποίο θα πολλαπλασιάζει το διοικητικό άχθος των επιστημονικών και ερευνητικών εργαστηρίων. Θα πρέπει να τεθεί αυτό το ερώτημα. Εγώ έχω επιφυλάξεις και συμμερίζομαι την ανησυχία των ερευνητών οι οποίοι φοβούνται ότι με ότι με τέτοιου είδους νομοθετήματα θα υπάρξει μεγάλη μεταφορά εγκεφάλων και ερευνητών γενικότερα σε άλλες χώρες με λιγότερο επαχθείς διοικητικές διαδικασίες. Ολοκληρώνω από εδώ Πρόεδρε λέγοντας ότι ε, θα πρέπει να απηχήσουμε τις ανησυχίες της κοινή γνώμης, ωστόσο φοβούμαι ότι η πρόταση της ε, Επιτροπής απομακρύνεται από τον θεμελιώδη στόχο της χρήσης των ζώων και θεμελιώδης στόχος της χρήσης των ε, ζώων σε πειράματα είναι να ενθαρρύνει την ε, πρόοδο της επιστήμης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Καπούλα Σάντος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι σήμερα στην Επιτροπή μας ε, καταφέραμε να δώσουμε το λόγο και στην κοινή γνώμη, όχι μόνο σε εμπειρογνώμονες ή σε ειδικού. Καταστήσαμε σαφές ότι μας ενδιαφέρουν ηθικά ζητήματα, μας ενδιαφέρουν θρησκευτικά ζητήματα, κοινωνικά, επιστημονικά. Δείξαμε ότι δεν είμαστε εθνοκεντρικοί, ε, δείξαμε ότι υιοθετούμε μία πολυπολιτισμική προσέγγιση. Και δείξαμε ότι δεν είμαστε εθνοκεντρική αλλά ούτε και υπερβολικά ανθρωποκεντρική. Έχουμε ευρύς ορίζοντες ένα ε, πολύ ανοιχτό πνεύμα αντίληψη των πραγμάτων και νομίζω ότι αυτό φάνηκε από όλες τις ε, ε, παρεμβάσεις των προσκεκλημένων μας. Δηλαδή στόχος μας είναι η επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ισορροπίας, της βέλτιστης δυνατής λύσης. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη σφαγή των ζώων, αναφέρομαι στο προηγούμενο θέμα, όμως μπορούμε να μεριμνήσουμε για τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες. Και στο θέμα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εξαλείψουμε την οδύνη ε, των ζώων τα οποία χρησιμοποιούνται σε πειράματα Μπορούμε όμως να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν λιγότερη οδύνη. Χωρίς τα πειράματα σε ζώα η ιατρική επιστήμη αυτή τη στιγμή θα είχε επιστρέψει στην εποχή ε, του χακού. Ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας. Ήταν πολύ χρήσιμες οι παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σανσορέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που είχαμε τη δυνατότητα κατά την ακρόαση να ακούσουμε τόσους εμπειρογνώμονες. Ο εισηγητής και πρόεδρος ε, της Επιτροπής μας ε, μπορεί, ε, ελπίζω να γράψει μια επιστολή που να συνοψίζει όλες τις θέσεις. Ακούσαμε τις παρεμβάσεις και είμαστε πεπισμένοι ότι τα πυρώματα σε ζώα και η χρήση των πρωτευόντων θηλαστικών δεν μπορούν να σταματήσουν τελείως. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να τα περιορίσουμε, θα πρέπει να θέσουμε ε, προϋποθέσεις, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε τελείως τα πειράματα σε ζώα, ούτε να σταματήσουμε τελείως τη χρήση πρωτευόντων θηλαστικών. Υπάρχουν και οικονομικές ε, πτυχές. Εάν ε, δεν συνεχίσουμε εμείς τα πειράματα στην Ευρώπη θα μεταφερθούν αλλού. Ακούστηκαν και άλλα επιχειρήματα. Δεν θα ήθελα όμως ε, να ε, ισχύουν, ε, να εφαρμόζονται μόνο οι οικονομικές, οι οικονομικοί συλλογισμοί στην έρευνα. Ακούσαμε πολλούς λόγους σήμερα γιατί δεν μπορούν να αποκλειστούν τα πειράματα σε ζώα. Κάθε πέντε χρόνια βλέπουμε σημαντικές πρόοδους στην ιατρική. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω και πάλι τη θέση. Ε, ότι ελπίζω κύριε Πρόεδρε ότι θα μπορέσετε να συντάξετε μια ε, ε, έκθεση η οποία να λέει ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τελείως τα πειράματα σε ζώα αλλά θα πρέπει να περιοριστεί στον βαθμό που είναι δυνατόν ε, η ταλαιπωρία των ζώων. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για το θέμα αυτό και όσο το εξετάζουμε κατά κάποιο τρόπο γίνεται και δυσκολότερο, αλλά αυτό που φάνηκε σαφέστατα είναι ότι υπάρχουν τμήματα της ε, σύστασης ε, των συστάσεων της Επιτροπής ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη το άρθρο 8 για παράδειγμα το άρθρο 10 για τα ζώα F2 είναι κάτι για το οποίο θα προτείνω να υπάρξει μια μελέτη εφικτότητας ε, ενός μιας τέτοιου είδους πολιτικής και σε, σε τι χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ σαφές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πήγαμε και στην Ελβετία να δούμε τι κάνουν οι Ελβετοί, γιατί οι Ελβετοί έχουν τρεις κατηγορίες σοβαρότητας ε, των ε, δοκιμών και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα καλό σύστημα. Θα το εξετάσουμε λοιπόν το άρθρο 45, οι εναλλακτικέ προσεγγίσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να ενισχύσω την εντολή του ΕΚΒΑΝ, του Ερευνητικού Κέντρου, να δούμε τι λύσεις υπάρχουν όταν Υπάρχουν εναλλακτικέ μέθοδοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία βέβαια ότι αν δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα ερευνητικά μας κέντρα, και δεν πρέπει να μας διαφεύγει βέβαια ότι και στα πανεπιστήμια γίνεται πολλή έρευνα, συχνά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι πρωτοστάτες αυτής της προσπάθειας, όταν δεν θέλω να βλέπω πειράματα σε ζώα, δεν θέλω βέβαια και η έρευνα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τότε τα πειράματα απλώ θα γίνονται υπό χειρότερε συνθήκε και ενδεχομένω ε, το αποτέλεσμα να μην είναι τόσο καλό. Νομίζω ότι αυτός, αυτή είναι η ισορροπία που προσπαθώ να επιτύχω. Θα δούμε βέβαια τις εναλλακτικές ε, επιλογές ε, όταν μπορούμε. Και πρέπει βέβαια να δούμε και την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, λεπτομερώς, γιατί πολύ συχνά μιλούμε και για την ε, κοινή γνώμη. Μπορεί βέβαια να υπάρξει και μία έρευνα που να λέει πιστεύετε στα πειράματα στη ζώα και η απάντηση θα είναι αρνητική, αλλά αν επίσης κάνουμε μία έρευνα που θα λέει δέχετε πειράματα, δέχεστε πειράματα σε ζώα εάν αυτό οδηγήσει σε φάρμακα που θα θεραπεύσουν ασθένειες. Η, η απάντηση θα ήταν μάλλον ναι. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ε, ξεύρουμε τη σωστή ισορροπία στην έκθεση αυτή. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό προσπαθώ να κάνω. Η ερώτηση που θα ήθελα να θέσω προς όλους τους εμπειρογνώμονες και νομίζω κύριε Μάτφιλτ εσείς μιλήσατε για την πολλή γραφειοκρατία είναι απαραίτητη η γραφειοκρατία όμως, ε, είναι δαπανηρή γραφειοκρατία ή είναι γραφειοκρατία για την οποία ε, θεωρείται ότι παρεμποδίζει ένα καλό σύστημα γιατί αν αυτή η τελευταία περίπτωση είναι η σωστή θα ήθελα να μου πείτε τι ιδέες έχετε ως προς αυτό. Αυτή είναι μια γενική ερώτηση που θέτω προς όλους τους εμπειρογνώμονες. Πώς εξασφαλίζουμε ότι ότι χρησιμοποιούνται οι εναλλακτικέ λύσεις, να είμαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούνται, ότι δεν είναι απλώς εμπόδια που ορθώνονται στις εναλλακτικέ αυτές επιλογές και πώς ε, ανταλλάσσουμε δεδομένα επιτυχώς. Γιατί Έχω κάποια δυσκολία ως προς το θέμα αυτό με τον κλάδο το φαρμακευτικό, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θέλετε να ε, ανταλλάσσετε πολλά από τα δεδομένα αυτά, αλλά αν πρόκειται να ε, επαναλαμβάνονται τα πειράματα χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, θα ήθελα να το ξέρω. Οπότε μπορείτε να μας πείτε ότι ε, θα ε, δεχθείτε ανταλλαγή δεδομένων με κάθε ειλικρίνεια. Γιατί δέχομαι τα πειράματα σε ζώα προς όφελος ανθρωπότητα, ανθρωπότητας, αλλά όχι διπλασιασμός των πειραμάτων, ώστε να διατηρήσετε τα πνευματικά δεδομένα ορισμένων ε, φαρμακευτικών εταιριών, γιατί ούτε αυτό μπορώ να τα αποδεχθώ. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θέλω να τα λάβω υπόψη, να τα ζυγίσω, για να καταλήξω σε μία έκθεση που πιστεύω ότι θα τύχει υποστήριξης στο τέλος και, νομίζω ότι από ηθικής απόψεως ε, έχω καταφέρει να βρω μια ισορροπία. Δεν είμαι πάντοτε, ε, δεν είμαι άνθρωπος που πάντοτε έχει ηθικά διλήμματα, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχω ένα πραγματικό ηθικό δίλημμα. και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά σας. Έχουμε ακόμη 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Αν μπορείτε να δευτερολογήσετε έκαστος για 4 λεπτά και μετά θα ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. Κύριε Μάτφιλντ, θέλετε να πάρετε το λόγο πρώτος. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα να πάρω το λόγο. Να πω καταρχάς ότι με ενθάρρυναν τα σχόλια τόσο τα δικά σας όσο και των άλλων μελών της Επιτροπής σας. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό, περίπλοκο. Ασχολούμαι με αυτό τα τελευταία 20 χρόνια. Ε, ψυχείτε και σώματι αν θέλετε κανείς ε, ε, θέλει να πάει και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη. Θέλει να πετύχει και τα δύο πράγματα μαζί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και να προστατεύσει τα ζώα. Και ενίοτε υπάρχει μια σύγκρουση δυσεπίλητη μεταξύ των δύο. Άρα ο μόνος δρόμος, η μόνη λύση είναι να υπάρχει σωστή ρύθμιση νομοθετική. Εμείς στα πανεπιστήμια αξιοποιούμε χρήματα από το δημόσιο κορβανά και συμφωνούμε απολύτως ε, να ξέρει η κοινή γνώμη τι κάνουμε με τα χρήματά τους και θα πρέπει όλα αυτά να απεικονίζονται στη σωστή νομοθεσία. Ε, δεν γίνεται καθόλου συζήτηση από αυτού. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Το θέμα είναι πώς επιτυγχάνονται όλα αυτά. Ε, με ρωτήσατε τι γίνεται με τη γραφειοκρατία όταν η νομοθετική ρύθμιση γίνεται τόσο επαχθής ώστε να αποτελεί τροχοπέδι για την επιστήμη. Κύριε Πρόεδρε, αναπόφευκτα οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει ένα εμπόδιο για την επιστήμη. Πάντοτε υπάρχει ένα τίμημα το οποίο καταβάλλεται. Το θέμα είναι άμα είναι το σωστό η οδηγία του 86 υλοποιήθηκε, εφαρμόστηκε με διάφορους τρόπους, ε, με αριστερά νομοθετήματα αλλά και με πιο ήπια νομοθετήματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μία από τις λίγες χώρες που θέσπισε άδειες για τα ιδρύματα, για τους ερευνητές και για την επιστήμη, για τους ε, επιστήμονες. Ήταν μία από τις λίγες χώρες στο Ηνωμένο Βασιλείο που υιοθέτησε αυτό το σύστημα των τριών επιπέδων αδειοδοτήσεων σε τρία επίπεδα. Πολλά παράπονα έγιναν ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές στο Ηνωμένο Βασίλειο διοργάνωσαν ακροάσεις όπου ακούστηκε αυτό το επιχείρημα ότι είναι πολύ πιο δίσκαμπτη η διαδικασία ώστε να διεξάγεται σωστή επιστημονική και πανεπιστημιακή έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκριτικά με άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία για παράδειγμα. Γνωρίζουμε όμως ότι αν ε, βρεθεί μια καινούρια ανακάλυψη ξαφνικά. Ε, δηλαδή, ένα γενετικό στροποποιημένο είδος ποντικού ε, και πει ο επιστήμονας ότι μπορώ να κάνω πείραμα στο συγκεκριμένο και να πετύχω πολύ σημαντικές ε, πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Ή θα ζητήσω ε, παράταση της άδειας και επέκταση της άδειας που έχω και θα χρειαστεί τρεις μήνες για να μου εγκριθεί ώστε να κάνω τον, ε, την έρευνά μου ή θα στείλω το μεταδιδακτορικό μου φοιτητή στην Καλιφόρνια να κάνει την ίδια έρευνα σε τρεις μέρες και να τη φέρει πίσω το αποτέλεσμα. Βλέπετε λοιπόν ότι Καλό είναι να υπάρχουν έλεγχοι, καλό είναι να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις έστω για να είναι σωστή η νομοθετική κάλυψη των ζητημάτων, αλλά στο βαθμό που χρειάζονται. Λένε πολλοί επιστήμονες ότι αν ακολουθήσω τους κανόνες, κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι είμαι βάναυσος ως προς τα ζώα. Θέλουμε κανόνες και ε, νόμους ώστε να κάνουμε πειράματα σε ζώα με το σωστό τρόπο. Και είναι σημαντικό αυτό για να αισθανόμαστε ασφάλεια και ανακούφιση και να μπορούμε να δουλέψουμε σωστά. Από εκεί και πέρα κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει η οδηγία αυτή να έχει διατάξεις οι οποίες να διευκολύνουν την πληροφόρηση για εναλλακτικές μεθόδους ερευνητικές. Όλοι θέλουμε να χρησιμοποιούμε ε, ερευνητικές μεθόδους που να προκαλούν όσο το λιγότερη ένταση ή οδύνη στα ζώα. Αν είναι γρηγορότερες οι μέθοδοι αυτές, αν είναι φθηνότερες, αν είναι καλύτερες, τόσο το καλύτερο για εμάς. Έχουμε επιστημονικά περιοδικά, έχουμε επιστημονικά συνέδρια. Είναι πολύ εύκολο να διαδίδονται αυτές οι πληροφορίες λοιπόν. Δεν υπάρχουν όμως οι ίδιοι διάβλοι, πληροφοριών για τις αναλλακτικέ μεθόδους. Θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρέπει να μας βοηθήσετε να τις γνωρίσουμε και να ακούμε για αυτές κάθε φορά που γίνονται. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φιλίπ Ντετιλέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στα αγγλικά όπως σας είπα και προηγουμένως. Όταν γίνεται λόγος για τη γραφειοκρατία, ε, θα ήθελα να πω το εξής. Βεβαίως και καλωσορίζουμε την νομοθεσία και πιστεύουμε ότι η οδηγία του 86 είναι απαξιωμένη, θα πρέπει να ε, αναθεωρηθεί και οι τωρινές διατάξεις θα βελτιώσουν την κατάσταση. Δηλαδή, θα έχουμε καλύτερη προστασία των ε, ζώων αλλά και των δικών μας δραστηριοτήτων. Θέλουμε σωστή λοιπόν νομοθετική ρύθμιση. ασκούμε κριτική σε όλες αυτές τις προστιθέμενες στιβάδες νομοθεσίας. Γιατί θα πρέπει να έχουμε αιτήσεις, αναθεωρήσεις και επανεξετάσεις όταν ήδη υπάρχουν τόσες πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν διετή αναθεώρηση και ότι προβλέπουν ότι φτάνει η διετής. Γιατί θα πρέπει να προστίθεται τώρα ετήσια. Γιατί μιλούμε για τη δημόσια περίληψη των ερευνητικών προγραμμάτων. Δεν το λέω για λόγους εμπιστευτικότητας, το λέω και για λόγους προστασίας των εργαζομένων μας. Στην εταιρεία μας, π.χ. στη Γερμανία, ε, ορισμένοι χημικοί επιστήμονες ε, υπέστησαν ε, διάφορες διώξεις όταν επέστρεφαν ε, στο σπίτι τους από διάφορους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων ακριβώς και μόνο επειδή το επώνυμό τους ήταν στην αίτηση για την απόκτηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ε, προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή θέλαμε να κινηθούμε. Αυτό ήταν το πνεύμα της παρέμβασής μας. Τώρα καταλαβαίνω ότι η μυστικότητα είναι κάτι το οποίο επιθυμούν οι εταιρείε για την επίτευξη συγκριτικού πλεονεκτήματος ή αυτό τουλάχιστον πιστεύουν οι υπόλοιποι για εμάς. Ωστόσο, δεν είναι ακριβώς ε, έτσι τα πράγματα. Κοιτάξτε την ε, πρωτοβουλία για την εναλλακτική ιατρική, κάτι το οποίο ήδη έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως. Οι εταιρείε ασχολούνται πάρα πολύ σε, με ερευνητικέ δραστηριότητε που έχουν να κάνουν με το Αλτσχάιμερ, με πάρα πολλά άλλα προβλήματα υγείας και συνεργάζονται μεταξύ τους. Βάσει του προγράμματος 6 έχουμε και toxmark Έχουμε ε, τα genomics. Έχουμε κατευθυντηρείς γραμμές, μοιραζόμαστε στοιχεία και πληροφορίες μεταξύ, των, μεταξύ μας. Ε, κάνουμε πειράματα πιστοποίησης της εγκυρότητας μαζί με την ΕΚΒΑΜ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο, το Αρμόδιο. Θέλουμε να μειώσουμε τα πειράματα στα ζώα ε, στην έρευνά μας για πάρα πολλές ασθένειες και πάρα πολλά προϊόντα. Στον τομέα της ασφάλειας μπορούμε να μοιραστούμε πολλές πληροφορίες μεταξύ μας χωρίς να τεθεί εν κινδύνο η ανταγωνιστικότητά μας. Και τελευταία παρατήρηση. Ε, τη δήλωση που έκανε για την Πέρτα και η οποία θα φύγει από την Ευρώπη. Οι εταιρείε υπόκεινται στους ίδιους κανόνες παντού στον κόσμο. Δεν μιλούμε μόνο για μελέτες και, μελέτες και δείκτες επιδόσεων. Μπορεί να υπάρχουν χώρες που λένε ότι μπορούν να μας προσφέρουν πρωτεύοντα θηλαστικά, όμως μπορεί εμείς να μην νομίζουμε ότι δεν έχουν αρκετή εχνηλασιμότητα ακόμα ή εγγυήσεις για τα ίδια αυτά. Είναι μακροπρόθεσμος όμως ο στόχος που ανέφερε προηγουμένως και θα πρέπει να επιδιωχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χόκενς. Είμαι επίσης δόκτωρ. Καταρχήν, θα ήθελα να απαντήσω στις παρατηρήσεις του κυρίου Άλιστερ. Με έκπληξή μου άκουσα ε, το πώς συνόψε τη δική μου ε, οδηγία, ε, ε την, πώς συνόψε τη δική μου ομιλία. δεν είμαι, πρώτη φορά με κατηγορούν για τόσο φαρατικές θέσεις, ποτέ δεν ήμουνα υπέρ μιας γενικής απαγόρευσης και θα απαντήσω τώρα στο ερώτημά σας, μην ανησυχείτε. θέλουμε περιορισμό της χρήσης των μη ανθρώπινων πρωτευόντων θηλαστικών. Ε, νομίζω ότι πρέπει να δεχτεί ο κόσμος ότι ε, ε, το σταμάτημα της χρήσης των πρωτευόντων είναι απόλυτα θεμητός στόχος και η χρήση των πρωτευόντων δεύτερης γενιάς είναι τρόπος να πετύχουμε την στρατηγική αυτή. Ε, εκφράστηκε η ανησυχία ότι ε, με την εφαρμογή τη οδηγία θα σταματήσουν όλες οι δοκιμέ σε ζώα στην Ευρώπη. Όχι θα σταματήσουν, θα αναγνωριστούν όμως τα ηθικά διλήμματα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι έχουμε οικογένειες, ε, όλοι ξέρουμε κόσμο που έχει υποφέρει, κόσμο που, περνά, που υποφέρει ακόμα. Τα ζώα υποφέρουν στι δοκιμέ. Γι' αυτό πρόκειται για δίλημα με την πραγματική έννοια του όρου. Ε, θέλουμε λοιπόν ένα ηθικό πλαίσιο ε, για να ε, για να εξετάζουμε την αναγκαιότητα και ε, την ε, ηθική του θέματος. Ε, τα τρία ρόη, αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση θα βοηθήσουν τους στόχους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έρευνα είναι απόλυτα ανταγωνιστική. Έχει το χρόνο και τα χρήματα να λάβει τις άδειε. Απλά το Υπουργείο Ιστορικών έχει εξετάσει το θέμα αυτό. Πολύ συχνά ο ερευνητής δεν έρχεται σε σωστή επαφή με τις αρχές ε, και αυτό είναι συνήθως το πιο ε, ρεαλιστικό σενάριο. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι μας θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κόσμος νοιάζεται για τις δοκιμές σε ζώα για πολύ καλούς λόγους. Δεν θα σταματήσουν οι δοκιμές, θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι θα σταματήσουμε ή να ζητήσουμε ή, να ε, ζητήσουμε απαγόρευση ε, οτιδήποτε ε, εκτός από τις πιο εξώφαλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, δηλαδή να ε, εξετάζονται κα, αποκλειστικά διακοσμητικά καλλιντικά σε ζώα. Όσον αφορά το μοίρασμα των δεδομένων, το Eurogroup πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την ΕΚΦΑΜ. Πέρα από αυτήν δεν υπάρχει συνεκτικότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επιστοποίηση των εναλλακτικών λύσεων και όπως ανέφερα και νωρίτερα είναι σημαντικό να εξετάσουμε όλο το ε, εύρος ε, των ε, δοκιμών. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις νέες τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιήσουμε όπου αυτό είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι ο Τζι μάλιστα αναφερόταν αποκλειστικά σε εσά. Ε, νομίζω ότι ήταν πιο γενικός, ε, ε, πολύ πιο γενική η παρατήρηση. Όχι, με, ανέφερε με συγκεκριμένο. α, καλά τότε. όχι, απάντησα στην παρατήρηση της ομιλήτριας ότι ήθελε πλήρη απαγόρευση για τα μεγάλα πρωτεύοντα και ότι θα πρέπει να ε, σταματήσει βαθμιαία η χρήση πρωτευόντων. Εντάξει, δεν θέλω να ε, ε, συνεχιστεί η συζήτηση. Αν θέλετε να επανέλθετε πολύ γρήγορα. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην απόλυτη απαγόρευση στα, στα μεγάλα πρωτεύοντα. Ήδη υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο μια εθελοντική ε, μείωση και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα με την απέτηση μιας ε, βαθμιαίας μείωσης της χρήσης των ε, πρωτευόντων. Ε, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε τη συζήτηση αυτή άλλο. Η κυρία Πετή Τζίμεν. Ε, ευχαριστώ πολύ. Όπως και η Δόκτωρ Χόκκινς θα ήθελα να απαντήσω σε μια παρατήρηση. Αναφέρθηκα στην αφέλεια. Και εγώ θα έλεγα μην κάνετε δοκιμές σε ζώα. Ε, όχι όμως αυτό, ε, δεν θα το έλεγα αυτό όμως αν αυτό σήμαινε ότι θα ε, τα μάτια μου ε, στον πόρο κάποιου ανθρώπου. Δεν θα έτρωγα τα ζώα, δεν θα τα κυνηγούσα, αλλά θα τα χρησιμοποιούσα σε δοκιμές αν ήταν απολύτως απαραίτητο. Όσον αφορά ε, συγκεκριμένα θέματα, η γραφειοκρατία. Κάποιες άλλες παρατηρήσεις ε, που έγιναν για την ομιλία μου ε, ήταν ε, ότι εκπροσωπώ την βιομηχανία. Η βιομηχανία πληρώνεται από τους αρρώστους και ερευνά για τους αρρώστους. Όσον αφορά τη γραφειοκρατία, η γραφειοκρατία πρέπει να είναι απαραίτητη, δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά επαχθής, ε, δεν θα πρέπει να εμποδίσει τη δημιουργία ενό ε, καλού συστήματος. Ε, πώς θα φροντίσουμε να μην εμποδίσουμε τη χρήση εναλλακτικών λύσεων. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με του νομοθέτες ώστε να φροντίσουμε τα πιστοποιημένα, οι εναλλακτικέ εναλλακτικές λύσεις να γίνουν χρυσά πρότυπα σε κάποιους τομείς. γίνεται πολύ καλή δουλειά στον τομέα των τριών ρόλων, αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση. οι δικέ μα φιλανθρωπικέ οργανώσεις ε, πρέπει να κάνουν έρευνες για τις διάφορες ασθένειες. Πρέπει όμως επίσης να συλλέγουν στοιχεία και να υποβάλουν εκθέσεις ε, σχετικά με εναλλακτικέ λύσεις. Υπάρχει εδώ ε, πολύ σημαντική τάση. Ε, αν τους δώσετε ε, μια λίρα για, να, για τις έρευνες για καρδιακές παθήσεις, απαιτούμε από αυτές να εξετάζουν την περίπτωση εναλλακτικών λύσεων. Όσον αφορά το μοίρασμα των δεδομένων, υπάρχει ε, μια διαμάχη στην ε, επιστημονική κοινότητα σχετικά με το θέμα της επικάλυψης των εργασιών και την... Ε, ε, απασχολεί πάρα πολύ συστηματική αναθεώρηση, δηλαδή συστηματική συλλογή όλων των ε, δεδομένων για ένα συγκεκριμένο θέμα που, ε, χρησιμοποιούνται πριν, που συλλέγονται πριν τις δοκιμές. Δεν γίνονται κλινικές δοκιμές εάν δεν, εξασφαλιστεί ποιος, εάν δεν διαπιστωθεί ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνουν οι δοκιμές αυτές. Εξετάζοντας τη δυνατότητα χρήσης των συστηματικών αναθεωρήσεων στις έρευνε σε ζώα. Δεν λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι δοκιμέ σε ζώα. Θέλουμε όμως σε κάθε βήμα να συλλέγονται όλα τα σχετικά και απαραίτητα στοιχεία ώστε να σταματήσει η ε, περιττή επανάληψη δοκιμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για τις ε, θέσεις σας ε, και τις ε, παρεμβάσεις σας. Αυτή τη στιγμή εκπονείται η έκθεση. Έχουμε προχωρήσει πολύ. Θα υπάρξουν αρκετές τροπολογίες και θα παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης στο Στρασβούργο στις 9 Μαρτίου. Θα έχουμε έτσι λίγες μέρες για να την τροποποιήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για τροποποίηση της ε, πρότασης ε, της ε, Κομισιόν, όχι απαραίτητα τη δική μου έκθεση, διότι το σχέδιο της έκθεσής μου ουσιαστικά αποτελεί σειρά τροποποιήσεων, τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής. Ε, κάναμε πολλή δουλειά για τις τροπολογίες αυτές, ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη έκθεση. Θα εξετάσουμε και τις ε, τροπολογίες που θα υποβληθούν και θα το αν ο συζητητής μπορεί να τις δεχτώ ή όχι. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ σήμερα. Ε, μπορέσαμε έτσι να έχουμε μια ισορροπημένη συζήτηση και να βρούμε έναν ε, τρόπο μπροστά στο θέμα αυτό. Θέλουμε οι δοκιμέ σε ζώα να γίνονται με τρόπο που να προστατεύονται τα ζώα ε, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. θέλουμε να γίνονται έρευνε, αλλά να χρησιμοποιούνται και εναλλακτικέ λύσει όπου υπάρχουν. Υπάρχουν ε, διαφωνίες ανάμεσα στην ε, βιομηχανία, τον, ε, τον πανεπιστημιακό κόσμο, τον ερευνητικό κόσμο και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την προστασία των ζώων, αλλά υπάρχουν και σημεία στα οποία συμφωνείτε. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσω να συμπεριλάβω όλα αυτά στην εκθεσή μου. Ελπίζουμε να έχουμε μια καλή έκθεση, διότι αλλιώς δεν θα περάσει από το Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ όλου, ευχαριστώ του βουλευτέ και του και τους, και τους, και τους, και Ευχαριστώ.